No,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

Cari colleghi, buonasera. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε και πάλι τη συνεδρίασή μα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Βόφραν αντιπρόεδρο της ε, Συνταγματικής Επιτροπής από το Εθνικό Συμβούλιο τη Αφιτερία. Κύριε έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί Εθνικοί Βουλευτέ, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτήν την ε, διακοινο... διακοινοβουλευτική συνεδρίαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ενώπιόν σα ω ε, εκπρόσωπο τη Συνταγματική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου τη Αυστρία ε, όπου θα σας ενημερώσω για την αυστριακή σκοπιά της ε, σημερινής μας ακρόασης. Η σωστή εφαρμογή και μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στο εθνικό δίκαιο είναι μια ουσιαστική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρησιμοποίηση του ενωσιακού δικαίου εξαρτάται κατά πολύ από την ε, μεταφορά του στο εθνικό δίκαιο, δηλαδή από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν ιδιαίτερη ευθύνη γι' αυτό. Ποιος ε, λοιπόν ο ρόλος ε, του Εθνικού Κοινοβουλίου. Καταρχά, είναι πολύ σημαντικό τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν την δυνατότητα να εξαντλήσουν όλες ε, τις ε, νομικές τους δυνατότητες ε, πριν και σε αυτό βοηθά πάρα πολύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Στο Σύνταγμα της Αυστρίας και στον εσωτερικό κανονικό του Κοινοβουλίου της Αυστρίας υπάρχουν διάφορα μέτρα για να ενισχύσουν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από το 1995 και την προσχώρηση της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε μέλος της ε, ομοσπονδιατής κυβέρνησης έχει ένα σύνδεσμο ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι σχέσεις έχουν ενισχυθεί. Υπάρχουν αιτιολογημένες ε, γνώμες οι οποίες πρέπει να καταρτίζονται ε, με βάση την αρχή της επικουρικότητας και εδώ να πω ότι η αρχή της επικουρικότητας είναι μία από τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας. Μέσω της αρχής αυτής ε, θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα μιας Ευρώπης που προστατεύει ε, μιας ενισχυμένης Ευρώπης ε, για τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίνει λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή και στα κράτη-μέλη ή τις ε, περιφέρειες που έχουν ανάγκη πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να έχουν αυτοδιάθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει κατά πολύ και ε, λογοδοτεί επίσης. Γι' αυτό όμως προϋποθέτει να ε, τηρούνται οι συνθήκες όχι σε όλους τους τομείς. Ε, ιδιαίτερα στην ε, ενιαία αγορά, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Νομοθεσία πρέπει να μεταφέρεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο Εθνικό Δίκαιο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία της. Επίσης, ε, η παράταση της ε, διαδικασίας κατάρτισης γνωμοδότησης στις 12 εβδομάδες είναι πάρα πολύ σημαντική. Το 2006 ενισχύθηκε ο πολιτικός ε, διάλογος και το αυστριακό, η Αυστριακή Βουλή, όπως γνωρίζετε, είναι χωρισμένη σε άνω και κάτω Βουλή και οι δύο έχουν σχέσεις με, ε, τους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ασχολούνται με ευρωπαϊκά ζητήματα και οι βουλευτές έχουν το καθήκον να ενημερώνουν τους πολίτες για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Εδώ το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο της Αυστρίας είναι το ε, πιο αρμόδιο και αυτό που έχει τις στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα όργανο το οποίο συνεισφέρει πολύ σημαντικά στην λειτουργία του κράτους, ε, διότι όχι μόνο συνδέει την κυβέρνηση με ε, τη, τα ομόσπονδα κρατήδια, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, οι σχέσεις ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό γίνεται μέσω των διαφόρων επιτροπών όπως η ΚΟΖΑΚ, η οποία την ε, περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε στη Βιέννη, αλλά και μέσω των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες. Με την ανταλλαγή αυτή απόψεων ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την εμπειρία των άλλων για να βελτιωθούμε. Το Κοινοβούλιο της ε, Αυστρίας χρησιμοποιεί διάφορα μέσα συνεργασίας με τις ε, Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά τις ε, ενωσιακές οδηγίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα συν ε, απόφασης και συνεισφοράς στο περιεχόμενο μιας οδηγίας, ας πούμε. Ε, επίσης, μπορούν να συνεισφέρουν έτσι ώστε μια οδηγία να γίνει κανονισμός. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, υπερθεματισμό, υπάρχουν ορισμένες εθνικές διατάξεις οι οποίες ε, προστατεύονται, αλλά υπάρχει, γίνεται μια ανάλυση έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ε, υπάρχει αυτός ο υπερθεματισμός. Επίσης, το έργο μας σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκτός από την ενημέρωση να γίνονται αναλύσεις, εξετάσεις ε, της νομοθεσίας σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στο δίκαιο, έτσι ώστε το έργο του Κοινοβουλίου να είναι αποτελεσματικό και πριν την έγκριση οποιασδήποτε ε, νομοθετικής πρότασης να έχουν αναλυθεί ενδελεχώς όλες οι πτυχές της ε, νομοθετικής πράξης. Η εκτελεστική εξουσία λοιπόν έχει πολύ σημαντικό έργο και Κοινοβούλιο κάτω και άνω βουλή συνεργάζονται άριστα, ασκούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο με όλες, τους τις ε, πτυχές, όλες τις Και τώρα, στα πλαίσια των λειτουργιών του Εθνικού Συμβουλίου της Αυστρίας υπάρχουν ειδικέ ομάδες αφιερωμένες στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις λέμε ώρες Ευρώπης μέλη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης δίνουν τακτικά αναφορά και ενημερώνουν για διάφορα ευρωπαϊκά ζητήματα και συμμετέχουν στις συνόδους κορυφής. Πολλές φορές μάλιστα βάζουν στην μερίσια διάταξη θέματα της επικαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωση που απασχολούν όλους. Οι Υπουργοί επίσης δέχονται ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της επαγγελματικότητας και οφείλουν να δίνουν απαντήσεις. Υπάρχει επίσης και μια επιτροπή αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιτροπή έχει άμεση και συνεχόμενη επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αυστρίας και τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει λοιπόν άμεση σύνδεση. Μετά, η ανταλλαγή απόψεων με ένα μέλος της ε, κυβέρνηση όχι μόνο διευκολύνεται αλλά και ασκείται τακτικά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ε, μεταφορά ε, του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο για να ασκείται έλεγχο ε, στην κυβέρνηση, αλλά και για να διαπιστώνεται η αποτελεσματική και γρήγορη μεταφορά της ε, ενωσιακή νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και προσβλέπω στην ε, γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέλτον. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το σημαντικό αυτό θέμα ε, που θα συζητήσουμε σήμερα. Οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, δίχως άλλο, θα μας δώσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο των δυσκολιών που αφορούν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από πολλαπλά επίπεδα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε απόλυτη συνείδηση της ύπραξης διαφόρων ε, προβλημάτων και αυτά οφείλονται στις εγγενείς διαφορές στο ε, ε, δικαστικά συστήματα που, και από άλλα θέματα λανθασμένη εφαρμογή, λανθασμένη μεταφορά χερνητικές αρνητικέ στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δημιουργεί αβεβαιότητες και εμποδίζει τους πολίτες και τους επιχειρηματίες να καρποθούν τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτη η εξασφάλιση όλων αυτών των στοιχείων αποτελεί προτεραιότητα. Το Κοινοβούλιο έχει μία σειρά από εργαλεία ελέγχου ελέγχου, όπως για παράδειγμα ε, προσωρινές ε, επιτροπές έρευνας για να διερευνηθούν περιπτώσεις κακοδιοίκησης ή παραβίασης, παραβάσεων. Αυτό αφορά όλου του πολιτικού κλάδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει και πολλέ αναφορέ από πλευρά των πολιτών. Πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να υιοθετήσει μια νομοθετική ε, ε, πρόταση ή να ξεκινήσει διαδικασίε επί παραλήψη κατά μια ε, χώρα μέλου. Κατόπιν πρόταση νομική επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή ένα ψήφισμα για την εφαρμογή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τελευταίο ψήφισμα της 14 η Ιουνίου 2018 το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για τον υψηλό αριθμό των επιπαραλήψεων διαδικασιών και αυτό μας δείχνει τη δυσκολία εξασφάλισης μια σωστή και άμεσης εφαρμογής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του δικαίου δεν είναι πρόσφατες και απαιτούν κοινέ προσπάθειες και στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Από την προπαρασκευή και την υιοθέτηση της νομοθεσίας ε, ε, και τον μετανομοθετικό έλεγχο και τη σωστή εφαρμογή. Η σημερινή συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και προκειμένου να έχουν μια άμεση και έγκαιρη συμμετοχή στον πολιτικό κύκλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρξει νομιμότητα και αποτελεσματικότητα και κατά συνέπεια αξιοπιστία των πολιτικών και των ε, ενωσιακών νομοθεσιών. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο ειδικού που θα έχουν 15 λεπτά στη διάθεσή τους για να παρουσιάσουν τις μελέτε τους. Θερμότητα την παράκληση να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευση. Θα πάρουν το λόγο μετά οι εκπρόσωποι του Ιταλικού, ε, Ελληνικού και Γερμανικού Κοινοβουλίου και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Βίμ Μπόλμα, ε, καθηγητή ε, Τη δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ε, dank. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Merci, danke, Ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Ε, τη δέχτηκα πολύ ευχαρίστως γιατί πραγματευόμαστε ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα σήμερα. Να σας πω λίγα λόγια. Καταρχήν είμαι εδώ για να σας κάνω μια ενημέρωση και μάλιστα σύντομη ενημέρωση γιατί λίγο χρόνο έχουμε και θέλω να μείνει χρόνος και για τη συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησαν ο κύριος Γκέρσλ και η κυρία Φεράρα με τη μεταφορά της ε, κοινωτικής νομοθεσίας σε εθνικό δίκαιο και τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία αυτής της μεταφοράς. Αν συζητούσαμε το ίδιο θέμα πριν από 40 χρόνια, θα ρωτήσω ένα πεντάλεπτο για τη συζήτηση. Γιατί τότε τα εθνικά κοινοβούλια δεν είχαν ιδιαίτερο ρόλο για τη μεταφορά στην εσωτερική ανομητάξη των κοινοτικών οδηγιών. Είχαν πολύ περιθωριακό ρόλο. Ελάχιστο λόγο είχαν στη θέση της κυβέρνησης του στο Συμβούλιο των Υπουργών και σίγουρα δεν ήταν στο επίκεντρο της διαδικασίας. Έκτοτε πάρα πολλά έχουν αλλάξει μέσα στα 40 χρόνια που πέρασαν. Εγώ βέβαια νομίζω ότι αν θα κουνούσα λίγο το μαγικό μου εργαλείο θα άλλαζαν οι διαφάνειες. Βλέπετε ότι πριν από 30 χρόνια τα εθνικά κοινοβούλια δεν ήταν ε, πλήρης ε, συνομοθέτες. Εξακολουθούν να μην είναι πλήρη συνομοθέτε για την κοινοτική, την ενωσιακή νομοθεσία. Έχουν έμεση επιρροή σε αυτήν, αλλά σίγουρα η επιρροή του έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν και από παραδοσιακή, παριθωριακή μάλλον και αδιόρατη θέση, πέρασαν να είναι ένα αναγνωρισμένο τρίτο μέρος και να εμπλέκονται ως τρίτο μέρος στις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχουμε πολιτικό διάλογο. Το είπαν και οι προλαλήσαντες. Επίσης έχουμε κάποια παραρτήματα στη συνθήκη της Λισαβόνας και το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Θα έρθω σε όλα αυτά τα σημεία αργότερα. Και πριν περάσουμε στην επίσημη ή ανεπίσημη άτυπη θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση τους στην Ευρωπαϊκή Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία, θα ήθελα να πω ότι η θέση των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων έχει αλλάξει. Ναι, μεν, αλλά με μεγάλες διαφορές. Έχουμε πραγματικά 27 πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους κόσμους. Τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ε, συνελεύσεις ε, ε, αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά εκεί σταματάν τα κοινά του σημεία. Έχουν περισσότερες διαφορές παρά κοινά σημεία τα διάφορα κοινοβούλια. Και μερικές φορές ακούω κάποιες πανικόβλητες φωνές, γιατί έχω δουλέψει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία 15 χρόνια. Ακούω λοιπόν κάποιε πανικόβλητε φωνέ για το τι κάνουν τα κοινοβούλια. Θα θυμάστε τη λευκή βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση το 2001, δεν κάνω λάθο. Που ξεκινούσε με δερμήτατη επίκριση του έργου των κρατών μελών και μάλιστα με πολύ βάσιμες μορφές γιατί όλε οι επιτυχίε όλες τις επιτυχίες σκαρπώνονταν τα κράτη-μέλη και όλε τι αποτυχίε τι τις επέριπταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Με αυτή την επίκριση ξεκινούσε η Λευκή Βίβλο. Και αυτό είναι άδικο εκ μέρους των κρατών μελών. Αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια ζουν στο δικό του κόσμο, στο δικό του πολιτικό κόσμο. Και αυτό δεν είναι από μόνο του κάτι αρνητικό αν του ρωτήσετε και είχατε το προνόμιο να πάρω συνεντεύξεις με πολλά μέλη κοινοβουλίων το 2006 και το 2009 από διάφορα κοινοβούλια, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, την Ιταλική Βουλή, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και διαπίστωσα ότι οι πολιτικοί και ιδιαίτερα οι κοινοβουλευτικοί έχουν την τάση να πιστεύουν ότι ο κόσμος γυρίζει ε, γύρω από αυτούς και ότι είναι το επίκεντρο του σύμπαντος και αν το κάνουν τη δουλειά τους έντοιμα, καλά κάνουν και το σκέφτονται, ότι έχουν την εξουσία να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξουν τον κόσμο, ότι ε, δικαιούνται να εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους τους και εκφέρουν τη φωνή των ψηφοφόρων τους. Όλα αυτά όμως έρχονται σε σύγκρουση με άλλους που έχουν την ίδια άποψη. Και αν το αναγάγουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε έχουμε μια εκτεταμένη πολιτική συζήτηση, που ούτε και αυτή από μόνη της είναι αρνητική. Τούτο λεχθέντος θα ήθελα να σταθώ λίγο στο τι κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και ποια είναι η θέση τους στην Ευρωπαϊκή Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία. Καταρχήν υπάρχουν διάφορα στάδια. Εγώ διέκρινα τρία. Καταρχήν, τα Εθνικά Κοινοβούλια διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην προετοιμασία της ε, ενωσιακής νομοθεσίας για τις οδηγίες για παράδειγμα, βέβαια δεν έχουν ρόλο στην έγκρισή τους, αλλά στη φάση της εφαρμογής και κυρίως στη φάση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο παίζουν ρόλο τα εθνικά κοινοβούλια. Πολύ συχνά μάλιστα παραβλέπονται στη φάση της αξιολόγησης. Εκεί παραμελούνται. Έχουμε διάφορες μελέτες και εκθέσεις τα τελευταία 15 χρόνια παντού στην Ευρώπη και ο καθηγητή Σμιθ, ο αγαπητό συνάδελφος, θα το σχολιάσει αυτό αργότερα φαντάζομαι, έχουν πρόβλημα με ένα κενό που υπάρχει στην, στο feedback για την ενωσιακή νομοθεσία, ιδιαίτερα όταν πάει κάτι στραβά στη διαδικασία της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Οπότε όταν κάτι πάει στραβά είναι λίγο δύσκολο να ληφθεί υπόψη και να τροποποιηθεί, γιατί θα πρέπει να επανέλθουμε στη διαδικασία της αναδιαπραγμάτευσης. Τα εθνικά κοινοβούλια από αυτήν την άποψη είναι πολύ σημαντικά, γιατί μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση, το τι συμβαίνει και να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου αν κάτι πάει στραβά και να στείλουν το μήνυμα στην κυβέρνηση προκειμένου αυτή να μεταφέρει το θέμα προς στο Συμβούλιο Υπουργών χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να ξεκινήσει νέα ή νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Οπότε το πρώτο στάδιο, το πρώτο σημαντικό τμήμα στο οποίο ενεργοποιούνται και παίζουν ρόλο τα, τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι σε ένα άτυπο στάδιο όταν υποβάλλεται η πρόταση για κοινοτική οδηγία στα κοινοβούλια και τους αποστέλλεται αυτή η πρόταση. Και αν θέλουν τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν κάποια επιρροή, τότε θα πρέπει να προλάβουν και αυτό το στάδιο. Γιατί αν περιμένουν να λάβουν πρώτα την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ήδη έχουν οριστικοποιηθεί κάποιες επιλογές Οπότε ήδη είναι κάπω αργά. Τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, που ακόμη συμμετέχει για τρει-τέσσερι μήνε ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μια πολιτική να προσπαθούν ε, να, εκφέρουν τη γνώμη τους ακόμη πιο νωρί στο στάδιο της δημοσίευσης πράσινης ή λευκής βίβλου. Και τότε ήδη να κοινοποιούν τη θέση της, ε, του Εθνικού Κοινοβουλίου προς την κυβέρνηση, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν την επίσημη υποβολή της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε πολλές περιπτώσεις τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια συμμετέχουν σε μια πρόταση κοινοτική οδηγίας, τη στιγμή που όμως τους αποστέλλεται ήδη η πρόταση. Και υπάρχουν διάφορα συστήματα α, για τη λήψη της πληροφόρησης Συνήθως υπάρχει ένα σύστημα διαλογής, συνήθως υπάρχουν μόνιμες επιτροπές παντού στην Ευρώπη, σε όλες τις ε, βουλές, που κάνουν την ε, διαλογή και λένε ότι αυτή η πρόταση είναι σημαντική, πρέπει να τη συζητήσουμε, ενώ η άλλη πρόταση δεν μας αφορά και πολύ. Οπότε γίνεται ένα σύστημα διαλογής ή προεπιλογής σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια και για τις σημαντικές ε, νομοθετικές προτάσεις ε, υποβάλλονται και κάποιες επιφυλάξεις ελέγχου. Γιατί ο το, η Βουλή κάνει πλήρη έλεγχο μιας πρότασης και μάλιστα τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλουν επιφύλαξη ελέγχου επιφύλαξη κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την κυβέρνησή του να σταματήσει, να διακόψει τι διαπραγματεύσει, να τι αναστείλει, μέχρι ότου το Κοινοβούλιο αποφανθεί επί τη προτάσεω. Και αυτό πριν από 12 χρόνια το φοβόταν πολύ, γιατί τότε μόνο η Δανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αυτή τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και μετά. Α, ε, απλώθηκε σαν πυρκαγιά παντού και όλοι άρχισαν να, να γύρουν επιφυλάξεις κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και τώρα είναι μανιτάρια. έχουν εμφανιστεί παντού αυτές οι επιφυλάξει του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και είναι ένα είδο φοβήτρου που χρησιμοποιούν τα κοινοβούλια και δεν το πολύ χρησιμοποιούν. Ο κύριος Γκέρσελ και η κυρία Φεράρα μας είπαν το πώς έχουν χρησιμοποιήσει τα κοινοβούλια τα μέσα για να επηρεάζουν τις κυβερνήσεις τους. Μπορούν να θέσουν ερωτήσεις, να εκδώσουν ψηφίσματα. Έχουν διάφορους μηχανισμούς τα εθνικά κοινοβούλια για να ασκήσουν επιρροή στην κυβέρνησή τους και να επηρεάσουν την θέση που θα λάβει η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών. Υπάρχουν όμως και κάποια νέα εργαλεία, νέοι μηχανισμοί. Έχουμε τον πολιτικό διάλογο, για παράδειγμα. Με βάση αυτό τον πολιτικό διάλογο, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να εκφέρουν τη γνώμη τους και ακόμη και η Μαλτέζικη Βουλή, η Βουλή ενός μικρού κράτους, σημαντικό με μικρό δεν, μπορούν να στείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Και από το 2006 έχουν υποβληθεί 5.000 ερωτήσεις και έχουν ε, δημοσιευτεί αντίστοιχε γνωμοδοτήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι καλό αυτό, γιατί τα λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι καλό αυτό για την ομοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα περάσω γρήγορα τις διαφάνειες. Έχουμε την ε, κίτρινη κάρτα, την πορτοκαλί κάρτα που προτάθηκε με, πολλούς, ε, με πολλές τυμπανοκρουσίες οι κίτρινες κάρτες χρησιμοποιήθηκαν μόνο τρεις φορές η διαδικασία αυτή. Συμβολικά έχει μεγάλη σημασία, κατοχυρώθηκε με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά στην πράξη δεν είναι και πολύ αποτελεσματική αυτή η διαδικασία. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να συντονίσει κανεί τι προσπάθειε μέσα σε 8 εβδομάδε όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων και να καταλήξουμε σε μια συντονισμένη θέση του ενός τρίτου τουλάχιστον των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και παρόλο που από πολιτική άποψη ε, έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Στην πράξη δεν πολύ χρησιμοποιήθηκε αυτή η διαδικασία, τρεις φορές μόνο. Ο πολιτικός διάλογος είναι ακόμη πιο σημαντικός μηχανισμός και λειτουργεί αρκετά καλά. Αυτό είναι το σημαντικό έργο και η ουσιαστική επιρροή που μπορούν να έχουν τα εθνικά κοινοβούλια στην φάση της διαπραγμάτευσης για μια νομοθετική πρόταση και όλο και περισσότερο πατάνε το πόδι τους στα εθνικά κοινοβούλια σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης με πολλούς και διάφορους τρόπους και αυτό είναι πολύ θετικό και θα το σχολιάσω αργότερα. Στη φάση της μεταφοράς, αυτό είναι πιο τεχνικό στοιχείο, εκεί τα Εθνικά Κοινοβούλια διδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών και η κυρία Φεράρα το σχολίασε για την Ιταλία, φυσικά και παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά οι σημαντικές επιλογές πολιτική έχουν ήδη γίνει Οπότε τα Εθνικά Κοινοβούλια απλώς είναι εκεί για να μεταφέρουν αυτές τις επιλογές στην ουσία ε, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην εσωτερική ένωμη τάξη, στο εσωτερικό δίκαιο. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτή η μεταφορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μεθόδους και τα εργαλεία που έχουν τα κοινοβούλια. Από το Σύνταγμα επίσης εξαρτάται, από τι μηχανισμούς δίνει το Σύνταγμα, γιατί μέσα δίνει το Σύνταγμα. Και βλέπουμε σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει ότι αν ένα εθνικό κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, στη διάρκεια της υποβολής της πρότασης, αν είχε συζητήσει το θέμα με την κυβέρνηση για την πρόταση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, τότε η μεταφορά είναι πολύ πιο εύκολη. Ένα κοινοβούλιο που έχει ευνηδιαστεί, που ξαφνικά του πέσε ορανοκατέβατη μια πρόταση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής φυσικά δεν θα βοηθήσει και πολύ, ούτε θα επιταχύνει τη διαδικασία τη μεταφορά. Οπότε όσο καλή προεργασία έχει γίνει, τόσο πιο γρήγορα γίνεται η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τα τεχνικά στοιχεία, βλέπουμε μεγάλη προτίμηση ε, για την δευτερογενή νομοθεσία και όχι την πρωτογενή. Όχι δηλαδή του Κοινοβουλίου. Αλλά αυτό φυσικά εξαρτάται από τα μέσα που προβλέπει το, κάθε σύνταγμα. Και φυσικά δεν είναι καμία φιλοσοφική λήθος. Το 2006 η ε, Ολλανδική κυβέρνηση μας έστειλε να κάνουμε περιοδία στην Ευρώπη και μας ενέθεσε να βρούμε ένα τρίκ, ένα τέχνασμα για να επιταχύνουμε τη μεταφορά. Γιατί τότε στον πίνακα επιδόσεων δεν είχαμε καλή θέση και έπρεπε να επιταχύνουμε την ε, μεταφορά βρίσκοντας ένα τέχνασμα ή αναζητώντας καλά παραδείγματα στη Δανία, Φιλανδία, Σουηδία και είδαμε πολλές καλές τεχνικές. Για παράδειγμα στην Ιταλία τότε είχαν ένα είδος ε, πολυνομοσχεδίου, omnibus. Ε, μία φορά το χρόνο είχαν ένα τέτοιο πολυνομοσχέδιο, omnibus, δεν θυμάμαι τον Ιταλικό όρο, οπότε μία φορά το χρόνο ε, με ένα πολυνομοσχέδιο μεταφέρονταν όλες οι οδηγίες. Στη Σλοβενία είχαν την διαδικασία fast track, εκτάκτο ανάγκης, Αυτά όλα φαινόταν καλά στα χαρτιά, αλλά στην πράξη δεν λειτουργούσε και πολύ, γιατί μία ε, ταχεία ε, μεταφορά προϋποθέτει δέσμευση και συμμετοχή σε προηγούμενα στάδια. Όταν γίνει καλή συμμετοχή και καλός έλεγχος, τότε θα είναι και γρήγορη η μεταφορά. Δεν είναι εδώ κανένα καμία φιλοσοφική λήθο. Πολλή συζήτηση γίνεται για τα τεχνικά θέματα. Αν θα πρέπει απλώς να γίνει απλή αντιγραφή ή να γίνει μια επεξεργασία ή ένας κανονιστικός υπερθεματισμός, το gold plating. Αυτό το είπε ο κύριο ε, Γκέρσλε. Αλλά όλα αυτά είναι λέξεις ε, αρκετά στομφώδεις, αλλά δεν γίνονται πολύ σπάνια. Στις κάτω χώρε ο κανονικός υπερθεματισμό των double banking ε, είναι σπάνια φαινόμενα. Και έρχομαι στα τελικά μου σχόλια, τα καταληκτικά. Θα έλεγε κανείς γιατί να έχουμε επικάλυψη με τα Εθνικά Κοινοβούλια, τις Εθνικές Κυβερνήσεις, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί να ενισχύσουμε τη θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Νομοθετική Διαδικασία. Το είπε καλύτερα ο Αλιμπράντι το 2018. Είπε ότι τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτή τη παρούσα φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουν ε, θεμελιώδη σημασία, γιατί η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο πολιτική, κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι θετικό. Γίνεται πολιτική συζήτηση, υπάρχει αντίλογος, αλλά Μία εξελιγμένη δημοκρατία χρειάζεται αντίλογο. Και αυτό γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λιμπράντι είπε λοιπόν ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν θεμελιώδη σημασία για την ομιμοποίηση τη ευρωπαϊκή πολιτική ή του ευρωπαϊκού πολιτικού βίου. Και γι' αυτό έχω μια ανησυχία που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σα. Και αφορά την επιτροπολογία. Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση εκχωρεί την, τις νομοθετικές της εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κοιτάξτε στα δεξιά Κοιτάξτε όμως το ανησυχητικό τμήμα, την κόκκινη πλευρά, το κόκκινο τμήμα, που αναφέρει το τμήμα της νομοθεσίας που εφαρμόζει ε, η Επιτροπή. Δεν είναι κατεξοδότηση πράξης του άρθρου 290 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλησαμε μετά την Λισαβόνα. Το Ευρωπαϊκό Κείμενο εξετάζει την κατεξοδότηση πράξη, αλλά περιθωριοποιήθηκε. Η κατεξοδότηση πράξης είναι κάτι που είναι σχεδόν σπάνιο. Το μεγαλύτερο τμήμα της επιτροπολογίας απορροφάται από τις εκτελεστικές πράξεις, τα εφαρμοστικά μέτρα που εμπίπτουν στο άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εμπειρογνώμονες. Και γι' αυτό προβληματίζονται και ανησυχούν και τα Εθνικά Κοινοβούλια και πολλοί πολίτες, γιατί πρόκειται για τεχνοκρατική, τεχνική νομοθεσία που εμπίπτει σε εκτελεστικές πράξεις και όχι στις κατεξιοδότηση. Βλέπω ότι αδειμονεί πρόεδρο και καλά κάνει γιατί έχω ξεντλήσει το τεταρτό μου. Ε, εν τα εθνικά κοινοβούλια αποκτούν όλο και σημαντικότερο ρόλο και πέρασαν από απλοί θεατέ ε, στο ρόλο του ενεργού παίκτη στη διαδικασία. Και αυτό είναι πολύ θετικό σε ό,τι αφορά τη ε, διαδικασία τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Επίση, ο μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση λειτουργεί, η διαδικασία με τι κάρτε ο πολιτικός ε, διάλογος λειτουργεί καλύτερα, γιατί για τις ε, κάρτες και τη διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίηση υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αλλά και τον πολιτικό διάλογο θα μπορούσαμε να τον αναπτύξουμε περαιτέρω. Και το πρώτο τελευταίο τμήμα, δεν υπάρχουν ε, θαυματούργε λύσεις για μια πιο γρήγορη μεταφορά. Πρέπει να αναμειγνύονται και να δεσμεύουν τα εθνικά κοινοβούλια. Μόνο έτσι θα εξασφαλίζεται ταχύτερη μεταφορά. Και ως προς την επιτροπολογία, η παλιού τύπου επιτροπολογία, ένα αντανακλαστικό πριν της Λισαβόνας 291 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μπούμεραν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ω διεθνού απολυτική οργάνωση. Κάτι που δεν ισχύει. Και ίσω θα πρέπει να τα μεταφέρουμε προ την άλλη πλευρά γιατί εκεί δεν έχουν έλεγχο οι Ευρωπαίοι πολίτε στι εκτελεστικέ πράξει. Αυτό θα ήταν μια πολύ κακή ιδέα, κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Μέλανη Σμιθ από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κάρτιβ. 15 λεπτά έχετε το λόγο. Uh, thank um, Σας ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη συνεδρίαση. Η παρουσίαση που θα σας κάνω αφορά τις ε, προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής ε, Νομοθεσίας, Ενωσιακής Νομοθεσίας στο Εθνικό Δίκαιο περιορίστηκα στις ε, διαδικασίες σε στην ε, παρουσίασή μου και γι' αυτό θα σας μιλήσω. Η έκθεσή μου αφορά επικαιροποιημένα στοιχεία για τις ε, περιπτώσεις παράβασης και θα σας δώσω μια συνοπτική εικόνα. Θα καλύψω λοιπόν σήμερα τρεις τομείς. Καταρχάς τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφαρμογή της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως μέρος της δέσμης μέτρων για την καλύτερη νομοθεσία. Περιλαμβάνει λοιπόν και την ε, πολιτική διαδικασία σε παραβάση. Συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη μου και ε, το 2018 με τα στατιστικά στοιχεία, αν και δεν είναι ακόμα επίσημα δημοσιοποιημένα. Και ε, να σταθώ σε κάτι που άκουσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το όργανο αρμόδιο με την για τη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Λοιπόν, αυτή η διαφάνεια μη σα τρομάζει, διότι αυτό που θέλει να πει είναι πολύ απλό. Όπως είπα, η πρόκληση που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτή, να κρατήσει για την Επιτροπή, να ελέγχει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου από τα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή οδηγίες ε, κτλ, αλλά και άλλα μέτρα εφαρμογής τα οποία λαμβάνονται από διάφορους ε, φορείς, τοπικού, τοπική αυτοδιοίκηση, ε, ή τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Όλο αυτό λοιπόν το διάγραμμα θέλει να περιγράψει τα στάδια στα οποία υπάρχει ρυθμιστική διαδικασία. Κάθε φορά δηλαδή που γίνεται παρέμβαση νομοθετική έχουμε την δυνατότητα παρέκκλησης από την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάθε ε, λοιπόν διαφάνεια είναι και μια ευκαιρία απομάκρυνση ε, από, τον ε, νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο δύσκολο να γίνει αποτελεσματική εφαρμογή του νοσιακού δικαίου. Ήθελα επίσης να αναφερθώ λίγο στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη νομοθεσία. Υπάρχουν μηχανισμοί στο άρθρο 258 διαδικασία επιπαραβάση και 216 οι οικονομικές κυρώσεις. Ε, όπως σας είπα θα σταθώ στη διαδικασία παραβάση. Τώρα, στο πλαίσιο της ε, ανακοίνωσης για την καλύτερη νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και άλλαξε προς ανατολισμό, επανακαθόρισε τον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα αυτό. Βασίζεται τώρα πλέον στους μηχανισμούς συμμόρφωσης. Δεν θέλει βέβαια να μειώσει τη σημασία των κυρώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάση. Όμως, όπως και να έχει, αυτό έχει επιπτώσεις ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, καθότι ε, είναι και νομοθέτης, αλλά και κρατά την Επιτροπή Υπόλογες και τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. Βλέπουμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές χρησιμοποιεί εκτελεστικούς κανονισμούς αφήνοντας έξω ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η καλύτερη νομοθεσία λοιπόν έχει στόχο ε, να απομακρυνθεί από την ε, συνήθινη νομοθετική διαδικασία και ε, περνά, κατευθύνεται περισσότερο στους εκτελεστικούς κανονισμούς της Κομισιόν. Η Κομισιόν δηλαδή είναι ο μόνος νομοθέτης σε ό,τι φορά του ε, μηχανισμού υποβολή εκθέσεων ε, τη Κομισιόν στην Επιτροπή Αναφορών και στην Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν προβλήματα στην πράξη διότι έχουν γίνει τρεις ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική επιβολής ε, της ε, Κομισιόν. Πρώτον, ανακοινώθηκε μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση ε, σε ό,τι φορά τις παραβάσεις. Δηλαδή, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον δεν θα ασκεί έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεως, αλλά σε αυτές που συμφωνούν με τις προτεραιότητές της. Έπειτα, το EU Pilot δεν θα χρησιμοποιείται πλέον. Σταδιακά εξελίφεται από το 2016 και αν δείτε την έκθεση του 2017 υπάρχουν ελάχιστες ε, υποθέσεις που ξεκίνησαν μέσω του EU Pilot μέχρι την σταδιακή εξάλληψή τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο προσπαθεί και έχει δαπανίσει πολλού πόρου ε, για την άντληση στοιχείων από τι εκθέσει αυτέ τη Κομισιόν. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει νέα σημασία στα μέτρα εφαρμογής με, τους, ε, με τα τακτικά αιτήματα για επιβολή κυρώσεων, κυρώσεων οικονομικών μέσω εμ, προστήμων που είναι κατά αποκοπή. Αυτές είναι οι κυριότερες αλλαγές λοιπόν που έχουν γίνει. Τώρα η παρουσίασή μου έχει πάρα πολλά γραφικά και πάρα πολλούς πίνακες. Αυτό που βλέπετε αφορά τις εκτίσεις εκθέσεις της Επιτροπής για τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τον συνολικό αριθμό διαδικασιών παραβάση που έχουν ξεκινήσει. Στην τελευταία εκθέση του Κοινοβουλίου φαίνεται πως έχουν μειωθεί αυτές οι διαδικασίες επί παραβάση, δηλαδή Μόνο 716 έχουν ξεκινήσει φέτος σε σχέση με τις 906 ε, πέρυσι. Αν δείτε όμως ε, τις τάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια θα δείτε ότι υπάρχει λίγο πολύ μια σταθερότητα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκινά 820 διαδικασίες σε παραβάση ανά κατά μέσο όρο και αυτή η διαφάνεια αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή σε πόσες ε, οδηγίες ε, φτάνουν στο στάδιο της εφαρμογής σε ένα δεδομένο έτος. Εάν δηλαδή υπάρχει μια πτώση του αριθμού των οδηγιών που πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο, υπάρχει και πτώση των ε, περιπτώσεων ε, διαδικασίας επί παραβάση. Αν αυξάνεται ο αριθμός των οδηγιών, αυξάνονται και οι διαδικασίες επί παραβάση. Οπότε βλέπουμε ότι η πτώση έχει άμεση σχέση με ε, τις διαδικασίες επί παραβάση. Υπάρχει, ας πούμε, μια πτώση 31% τελευταίο έτος. Σε γενικές γραμμές λοιπόν παρατηρείται μια σταθερότητα στην ε, κίνηση νέων διαδικασιών παραβάση. Τώρα, όσον αφορά τι τάσει των τελευταίων ε, πέντε ετών, νομίζω πως όπως ε, είδαμε και από την περίπτωση του περιβάλλοντος το πρωί, το περιβάλλον είναι ο κύριος λόγος κίνησης διαδικασίας σε Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών το 17.864 ε, καταγγελίες. Το περιβάλλον ήταν στην δεύτερη θέση. Επίσης, το περιβάλλον είχε τις περισσότερες υποθέσεις ε, που ξεκίνησαν μέσω του EU Pilot και η δεύτερη διαφάνεια δείχνει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια και σε γενικές γραμμές τα τελευταία 20 χρόνια το περιβάλλον είναι πρώτο σε αριθμό καταγγελιών ακολουθείται στενά από τις μεταφορές και τις δημοσιονομικές υποθέσεις, δημοσιονομική σταθερότητα. Σε ό,τι αφορά τις ε, περιπτώσεις, τις υποθέσεις τις οποίες η Κομισιόν παρέπεμψε στο δικαστήριο το 2017, 28 ε, υποθέσεις ε, παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο και πάλι το περιβάλλον στην πρώτη θέση, εσωτερική αγορά και δικαιοσύνη. Και λυπάμαι τα γράμματα είναι πάρα πολύ ε, μικρά. Ε, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Πολωνία ήταν ε, οι χώρες με τις περισσότερες τέτοιες υποθέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικαστικές αποφάσεις, το δικαστήριο εξέδωσε 16 αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 258. Οι χώρες με τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις ήταν η Γερμανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Οι, κύριοι, οι κυριότεροι τρει τομεί ήταν πάλι περιβάλλον, φορολογία και μεταφορέ. Μία ε, απόφαση επίση ε, αφορούσε το άρθρο 262, οικονομικέ κυρώσει ε, κατά τη Ισπανία για μία υπόθεση ελευθερία εγκατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες ξεκινούν από διαδικασία παραβάση, περνάνε στο δικαστήριο, βλέπουμε ότι υπάρχουν τάσεις ε, στον τύπο των υποθέσεων, το περιβάλλον στην πρώτη θέση, οι μεταφορές σε δεύτερες και παρά το γεγονό ότι η Κομισιόν χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία για συμμόρφωση, για παράδειγμα την έκθεση εφαρμογή ε, τη ε, Κομισιόν, διαφορε εκδηλωσει διάφορα εργαστήρια, παραμένει το πρόβλημα. Επίση. το οι μεταφορές ε, εξακολουθούν να είναι πολύ ορατές και έντονα παρούσες στην όλη διαδικασία. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια όμως, μετά το περιβάλλον, τη φορολογία και την δημοσιονομική σταθερότητα, αρχίζουν και εμφανίζονται νέοι τομείς. Αυτά λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία συμφωνούν και με αυτά που μαθαίνουμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τι φραγμούς ε, αυτά αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς ε, του δικαίου που είναι πάρα πολύ περίπλοκοι, περιβάλλον, ε, δημοσιονομικοί κανονισμοί, φορολογία. Υπάρχουν μετά τομείς οι οποίοι είναι αρκετά αφορούν ζητήματα αρκετά λεπτά και ευαίσθητα για ορισμένα κρατημέλη και εκεί εντοπίζονται οι δυσκολίες. Αυτά λοιπόν είναι τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα άμεσα και δημόσια. Έχω χρησιμοποιήσει και άλλα στατιστικά στοιχεία τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α πούμε, δεν θα δημοσιεύσει τα επόμενα στοιχεία για τις διαδικασίε σε παραβάση μέχρι τον Ιούλιο του 2019, αλλά έχω κάποια στοιχεία μέχρι τον Οκτώβριο και τον Οκτώβριο του 2018 και βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι τις 17 Οκτωβρίου υπήρξαν 27 υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο. Πέρυσι μόνο 28 συνολικά ήταν οι υποθέσεις. Και οι τρεις κυριότεροι τομείς των υποθέσεων αυτών ήταν περιβάλλον, μεταφορές, ενέργεια. Και όπως βλέπετε υπάρχει μία σημαντική αύξηση σε περιβαλλοντικές καταγγελίες. Ε, για όλο το 2017 λοιπόν είχαμε μόνο 16 ε, περιβαλλοντικές υποθέσεις που αρπέμφθηκαν στο δικαστήριο. Ενώ τώρα έχει αλλάξει ο αριθμό αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι οικονομικέ κυρώσει, υπήρξε μια καταδικαστική απόφαση κατά τη Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 262 για το περιβάλλον, και μια ε, περίπτωση οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθη από το δικαστήριο φέτο κατά τη Ελλάδα και πάλι για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Όπως ε, είπα λοιπόν, όταν ετοίμαζα την ενημέρωση και την παρουσίαση αυτή, έκανα μία έρευνα ε, και στα Εθνικά Κοινοβούλια και οι εκθέσεις ε, εκεί επισημαίνουν 10 τομεί που βρήκα και στην ερευνά μου, οι οποίοι συνεισφέρουν στην δημιουργία εμποδίων στην εφαρμογή του νοσιακού δικαίου. Από αυτού τους 10 τομεί, μόνο τρει είναι υπό τον έμεσο έλεγχο των θεσμικών οργάνων η χαμηλή, ο χαμηλό, ο μη περίπλοκος χαρακτήρας. Δηλαδή, όσο πιο απλή είναι η νομοθεσία, τόσο καλύτερη η εφαρμογή. Και αυτό φυσικά είναι ε, ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σχεδιάσει μια απλή νομοθεσία, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ε, ολοκληρώσει την νομοθετική διαδικασία. Η εφαρμογή λοιπόν του νοσιακού δικαίου θα πρέπει να είναι ευθύ εξ αρχή στο νου του νομοθέτη. Έπειτα, το δεύτερο εμπόδιο είναι η εθνική ε, ικανότητα επιβολής και ο έλεγχος. Όσο περισσότερη η γραφειοκρατία, τόσο δυσκολότερη η εφαρμογή. Αυτό είναι ζωτική σημασίας για να διαπιστώσουμε και να διασφαλίσουμε μάλλον ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα μεταφέρεται στην εθνική. Επίσης υπάρχουν διάφορα, διάφορες ε, προτάσεις ε, κατάρτισης ε, του δικαστικού προσωπικού των αρχών επιβολής του νόμου. Τέλος, ο τρίτος παράγοντας είναι η, είναι η εφαρμογή και ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των θεσμικών οργάνων. Εδώ το Κοινοβούλιο έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως φαντάζεστε, και διότι αποτελεί βήμα για τους πολίτες να εκφράσουν ε, τη δυσαρέσκειά τους, τα παράπονά τους, αλλά και επειδή είναι το θεσμικό όργανο στο οποίο λογοδοτεί η Επιτροπή. Κλείνοντα λοιπόν, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τον μηχανισμό υποβολή εκθέσεων ε, τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση τη Κομισιόν. Ε, είναι πολύ σημαντική έκθεση, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, ε, διότι ακριβώς σε αυτό λογοδοτεί η Κομισιόν. Αναλύοντας λοιπόν την έκθεση και τις εκθέσεις μάλλον τα τελευταία δέκα χρόνια, παρατηρούμε, αν κάνουμε μία ανάλυση κατά τομέα, ότι υπάρχει μία ιεράρχηση και βλέπουμε πόσο χρόνο δαπανάει η Επιτροπή για ποια θέματα. Βλέπουμε ότι ξεχωρίζουν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Το Κοινοβούλιο λοιπόν μέσω της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ε, συζητά τα επίγοντα ζητήματα και φυσικό αυτό διότι είναι πολιτικό όργανο, όμως τα ε, επίγοντα ζητήματα δεν έχουν πολλές φορές να κάνουν ούτε με την ε, αποτελεσματική εφαρμογή του ανασιακού δικαίου, ούτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διαδικασία ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επίσης ε, υπάρχει και θέμα με την διαφάνεια των ε, δεδομένων σχετικά με, την, με τις Τώρα, πολύ χαμηλά στη λίστα βρίσκεται ε, η νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο προσέχει πάρα πολύ να δίνει την ε, δεούσα προσοχή στην ε, καλύτερη νομοθεσία και τις ε, νέες πρωτοβουλίες. Διότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απομακρύνεται από τις κυρώσεις και κατευθύνεται προς μηχανισμούς συμμόρφωσης, τότε ο έλεγχος της Κομισιόν αφορά και τον έλεγχο αυτών των πρωτοβουλειών. Για παράδειγμα, τι ποσοτικά και ποιοτικά κάνει η ε, έκθεση εφαρμογής, που, πώς συνεισφέρουν αυτοί οι μηχανισμοί στην, ε, στον αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξοδεύει κονδύλια για αυτούς τους μηχανισμούς, πρέπει να ελέγξουμε αν αυτή είναι αποτελεσματική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι σταδιακά καταργείται ε, το EU Pilot. Αυτά λοιπόν εν συντομία ε, τα σχόλιά μου για την εκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ξεκινάμε με τον κύριο Ρωσίνη. Για 10 λεπτά εκπροσωπεί η κυρία Ρωσίνη, εκπροσωπεί το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά μας για να μιλήσουμε μεταξύ κοινοβουλίων και να δούμε πώς τα κοινοβούλια συνεργάζονται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η δραστηριότητα του Ιταλικού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναδιαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και αυτό μετά από μία μεταρρύθμιση η οποία έγινε το 2012 με το νόμο 234 που επαναδιοργάνωσε την όλη διαδικασία στην ουσία χωρίζοντας ένα νόμο σε δύο νομοθετικές διατάξεις, δύο διαφορετικοί νόμοι δηλαδή προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια προσαρμογή μεταξύ των άλλων του συστήματός μας. Αυτές οι δύο ξεχωρικές διατάξεις είναι ο νόμος εξουσιοδότησης που περιέχει διατάξεις εξουσιοδότησης στην κυβέρνηση που είναι αναγκαίες προκειμένου να γίνουν δεκτές οι κοινοτικές οδηγίες και ο ευρωπαϊκός νόμος ο οποίος εγγυάται απευθείας τη συμμόρφωση του Ιταλικού, της Ιταλικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή. Για ποιο λόγο αυτή η μεταρρύθμιση. Γιατί στο παρελθόν Βρεθήκαμε ενώπιον ενός διεξόδου λόγω της μη έγκρισης ορισμένων διατάξεων που περιείχαν τα κοινοτικά σχέδια νόμου και τα οποία είχαν δημιουργήσει προσκόμματα στην εφαρμογή του νόμου και την έγκριση του νόμου. Σκεφτήκαμε λοιπόν να χωρίσουμε στα δύο αυτό το μέσο και αυτό για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ταχύτητα προσαρμογή στα κοινοτικά δεδομένα και από την άλλη πλευρά προκειμένου να αποκλείσουμε την ένταξη στα ευρωπαϊκά σχέδια νόμου ξένων θεμάτων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια έγκαιρη προσαρμογή από μέρους του Ιταλικού, της Ιταλικής νομοθεσίας. Τι περιέχουν ε, συντομία οι δύο αυτοί νόμοι. Ο νόμος Ευρωπαϊκής Εξουσιοδότησης περιέχει εξουσιοδοτήσεις στην κυβέρνηση για την εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων. Περιέχει επίσης τον όλο μηχανισμό κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων και περιέχει και τις σημαντικές αρχές για θέματα για τα οποία είναι αρμόδιες οι περιφέρειες. Ο νόμος ε, ε, ευρωπαϊκής ε, εξουσιοδότησης ορίζει τα βασικά κριτήρια και τις αρχές εξουσιοδότησης με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί η κυβέρνηση και εισαγάγει και την απαγόρευση του αποκαλούμενου gold plating, δηλαδή απαγόρευση του να υιοθετηθεί μία πιο περιοριστική νομοθεσία σε σχέση με την απαιτούμενη από τις ίδιες τις οδηγίες. Ο ε, νόμος Ευρωπαϊκής Εξοδότησης μπορεί να εισαγάγει συγκεκριμένες αρχές και κριτήρια επιπροσθέτως κριτήρια τα οποία η κυβέρνηση θα πρέπει να σεβαστεί. Στον Ευρωπαϊκό Νόμο, το δεύτερο μέσο, περιέχονται οι κανόνες άμεσης εφαρμογής που στόχο έχουν την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που αποτε και αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών προ ε, παραβίες και παραβίες. Δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Νόμος τακτοποιεί τα πράγματα εκεί που η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει το βάσιμο των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιέχει επίσης κανόνες προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοστούν διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναυτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει ως έχει η δυνατότητα της κυβέρνησης να υιοθετήσει κατεπήγοντα μεταξύ των άλλων μέτρα διαφορετικά από αυτούς τους δύο νόμους σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο προκειμένου να ε, αντιμετωπιστούν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Η όλη κοινοβουλευτική διαδικασία προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά σχέδια νόμου ευρωπαϊκής εξουσιοδότησης εξετάζονται σε μια ειδική ευρωπαϊκή ολομέλεια που ε, συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν όλες οι μόνιμες επιτροπές του Εθνικού Κοινοβουλίου. Στην ε, Βουλή η εξέταση αυτή γίνεται στην Επιτροπή Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκω και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας στις 13 μόνιμες επιτροπές. Πού οδήγησε αυτή η μεταρρύθμιση του 2012 κατέστησε πιο αποτελεσματική όλη τη φάση εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών στο Ιταλικό, στην Ιταλική νομοθεσία. Στα προηγούμενα πρώτα χρόνια η μεταρρύθμιση χρησιμοποιήθηκε οδηγώντας στην έγκριση ε, κάθε νόμο των δύο νόμων ευρωπαϊκής εξουσιοδότησης. Μέση διάρκεια των εργασιών 5 έως 6 μήνες που το κάθε χρόνο για την εξέταση και την οριστική έγκριση των δύο νόμων. Με αυτόν τον τρόπο, τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια το Ιταλικό Κοινοβούλιο μπόρεσε να εξασφαλίσει ακρίβεια και ταχύτητα στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων σε κάθε έτος αναφοράς. Σε αυτή την νομοθετική περίοδο θα ήθελα να θυμίσω ότι μόλις εγκρίναμε το σχέδιο νόμου Ευρωπαϊκής Εξουσιοδότησης που έχω μαζί μου το εγκρίναμε πριν από δύο εβδομάδες. Αυτές τις μέρες είναι υπό ε, ε, εξέταση στην Γερουσία όπου συζητείται και ο δεύτερος νόμος, ο ευρωπαϊκός νόμος που θα περάσει μετά σε μάσα στην Βουλή. Μέχρι το τέλος του χρόνου το Ιταλικό Κοινοβούλιο θα ολοκληρώσει με την έγκριση των δύο νόμων που αποτελούν την καρδιά της δραστηριότητας ε, μεταφοράς και εφαρμογής στο εθνικό ε, δίκαιο. Ποιες είναι οι άλλες θετικές επιπτώσεις αυτής της μεταρρύθμισης η βελτίωση που προέκυψε ως προς τις διαφορές που έχουν σχέση με την Ιταλία. Ιδιαίτερα την περίοδο 2014-2018 ε, οι διαδικασίες ε, επί παραβάση από 121 μία πέραστα στις 68 εκ, των οποίων 60 για παραβίαση του ε, ενωσιακού δικαίου και 8 για ελλειπή μεταφορά οδηγιών. Η μεταρρύθμιση του 2012 σήμαινε ότι το, Ιταλικό Κοινοβούλιο ασκεί απόλυτο έλεγχο στις διαδικασίες επί Η κυβέρνηση καλείται να, ε, ε, λογοδοτήσει στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κάθε τρεις μήνες ενημερώνει το Κοινοβούλιο και κάθε έξι μήνες ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις οικονομικού χαρακτήρα. Πέραν αυτού θα πρέπει να αιτιολογήσει στο Κοινοβούλιο τις ε, ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη μεταφορά στο εθνικό ε, δίκιο ανακοινώνει στην κυβέρνηση και στο κοινοπούλιο την πορεία των διαδικασιών επί παραβάση και ενημερώνει για κάθε σημαντική εξέλιξη που να τις αφορά. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει μια διαδικασία για την εξέταση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από πλευράς των αρμόδιων μόνιμων αρμόδιων επιτροπών, οι οποίες μπορούν να εκφέρουν την άποψή τους στην κυβέρνηση ως προς την ανάγκη λήψης πληροφοριών, ε, ε από πλευράς της κυβέρνησης με αναφορά στα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Θα θέλαμε να πούμε ότι όλοι οι Ιταλικοί νόμοι προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση μεταξύ των τελικών νόμων και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποτελούν αντικείμενο διαρκούς εξέτασης από πλευράς της Επιτροπής μου, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Πολιτικών που διαβιβάζει τη γνωμοδότησή του σε όλες τις μόνιμες επιτροπές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την γνωμοδότηση στα πλαίσια των νομοθετικών τους ε, ε, ερευνών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, κυρία Ρωσίνη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, τον κύριο Σαρακιώτη, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Σαρακιώτη, παρακαλώ, για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> ξεκινώντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τι δύο συνδιοργανώτριε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μα έδωσαν την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει και κυρίω να ενημερωθούμε για τι βέλτιστε πρακτικέ άλλων κοινοβουλίων για ένα θέμα τόσο σημαντικό όπως αυτό που εξετάζουμε σήμερα. Για τη Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε διατάξεις του κανονισμού μας σχετικές με τον έλεγχο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τόσο εξάντε όσο και εξπόστ, οπότε η συνάντηση αυτή αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία να αποκομίσουμε νέες ιδέες και να εξετάσουμε αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά με στόχο πάντα τη βελτίωση της νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Το βάρος της διαδικασίας ενσωμάτωσης έχει η κυβέρνηση και η Ελληνική Βουλή ψηφίζει τα νομοσχέδια που αφορούν μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Ειδικά Όσον αφορά το σκέλος της εφαρμογής, θα πρέπει να επισημάνω ότι η εμπειρία του Κοινοβουλίου μας στον τομέα αυτό είναι μικρή. Ωστόσο υπάρχουν διάφορες ιδέες που θα θέλαμε να υλοποιήσουμε προκειμένου να διαμορφωθεί στη συνέχεια και το ανάλογο κανονιστικό πλαίσιο. Αρχικά θα ήθελα να περιγράψω εν συντομία τα στάδια που ακολουθούνται στη χώρα μου από τη στιγμή της δημοσίευσης μιας νομοθετικής πρότασης μέχρι την υιοθέτησή της και τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώνει δια των εκπροσώπων της τα καθήλυνα αρμόδια Υπουργεία με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στο Υπουργείο Εξωτερικών περί των κυοφορουμένων πρωτοβουλειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εθνική αντι... Οι εθνικοί εκπρόσωποι διαπραγματεύονται ανάλογα στις ομάδες εργασίας και στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, μπορεί η Βουλή μέσω των επιτροπών της να συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην εξοικείωση των βουλευτών με θέματα που θα τους απασχολήσουν στο μέλλον, είτε στο στάδιο ελέγχου επικουρικότητας ή στο στάδιο της ψήφισης νομοσχεδίου ενσωμάτωσης, αλλά και στη συνδιαμόρφωση εθνικής θέσης, γεγονός το οποίο διευκολύνει και το έργο των αρμοδίων χειριστών των Υπουργείων και της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας που συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές ομάδες εργασίας. Κατά την πρώτη εβδομάδα από τη δημοσίευση σχεδίου νομοθετικής πράξης και τη διαβίβαση στη Βουλή των σχετικών εγγράφων από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίνει σε εφαρμογή η εσωτερική διαδικασία που οδηγεί σε παραπομπή ή μη της πρότασης σε έλεγχο επικουρικότητας από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και τις καθήλυν συναρμόδιες επιτροπές. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει την πορεία των πραγμάτων ως προς την αρχή της αναλογικότητας μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, του πολιτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διατύπωση απλής γνώμης, της συνεργασίας με τις αντίστοιχες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκληθούν να εξετάσουν τις νομοθετικές αυτές προτάσεις και της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας εν γέννη το νομικό τμήμα της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει την έκδοση σχεδίου οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωση στο οικείο Υπουργείο, το οποίο θα αναλάβει την επίσπευση της διαδικασίας ενσωμάτωσης. Κοινοποιεί επίση σε συναρμόδια Υπουργεία, στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνηση καθώς και στην Ειδική Νομική Υπηρεσία. Συγχρόνως, το Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ζητά από το Επισπεύδον Υπουργείο αρχικό πλάνο ενσωμάτωσης, το οποίο περιλαμβάνει ενημέρωση ως προς το χρονοδιάγραμμα, τις αρμοδιότητες, τυχόν αντικρουόμενες υφιστάμενες διατάξεις και άλλα. Το επισπεύδον τώρα Υπουργείο γνωστοποιεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και κοινοποιεί στην Ειδική Νομική Υπηρεσία και την μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πλάνο ενσωμάτωσης. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης παρέχει υποστήριξη στα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία εν συνεχεία ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία για τυχόν τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος το εθνικό μέτρο μεταφοράς, είτε ο νόμος, είτε προεδρικό διάταγμα, είτε υπουργική απόφαση, θεωρείται από τον Γενικό Γραμματέα κατόπιν ελέγχου από το Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων σε συνεργασία με το Νομικό Γραφείο. Το Εθνικό Μέτρο Μεταφοράς δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Το Γραφείο Συντονισμού, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Υπουργείο, ενημερώνει την ειδική νομική υπηρεσία και το νομικό τμήμα της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας για τη δημοσίευση της πράξης ενσωμάτωσης. Ε, η ειδική νομική υπηρεσία κοινοποιεί το Εθνικό Μέτρο Μεταφοράς που υιοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ειδική ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η Επιτροπή κατόπιν εξιοδότησης της ελληνικής δημοκρατίας το αναρτά στο Eurlex η Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαμορφώνει σε αιτήσια βάση πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, στην οποία αποτυπώνεται η επίδοση των κρατών μελών, διαμορφώνεται ο ενωσιακός μέσος όρος και τίθεται ο στόχος για το ανώτατο έλλειμμα μεταφοράς. Στον πίνακα επιδόσεων εσωτερικής αγοράς του 2017, η Ελλάδα εμφανίζει 0,9% έλλειμμα ενσωμάτωσης, με στόχο 1% και μέσο όρο ευρωπαϊκό 1,5% και κατατάσσεται 8η μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ο εκτιμόμενος δείκτης συμμόρφωσης των υιοθετούμενων από την Ελλάδα εθνικών μέτρων μεταφοράς προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 0,2%, με στόχο 0,5% και μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0,6%. Ε, η χώρα μου βρίσκεται στα έξι κράτη-μέλη με τις λιγότερες πλημελώς ενσωματωμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι σταθερός στόχος της Ελλάδος είναι το έλλειμμα ενσωμάτωσης οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κατώτερο του 1% σύμφωνα και με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελών το 2007. Παραμένει επίσης στόχος οι συγκεκριμένες επιδόσεις της χώρας να έχουν σταθερότητα και συνέχεια χωρίς σε καμία περίπτωση να παραβλέπεται η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας της εθνικής μας νομοθεσίας όταν θεσπίζεται σε συμμόρφωση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό αποτελεί μέλημα η έγκαιρη ενσωμάτωση να συνοδεύεται από μια πολύ προσεκτική επιλογή του μέσου ενσωμάτωσης. Η διασφάλιση της δυνατότητας απρόσκοπτης εφαρμογής του εθνικού δικαίου, αλλά και ανάλογη προσαρμογή των διοικητικών διαδικασιών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την υποστήριξη εφαρμογής της νέας νομοθεσίας η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει μέχρι τώρα ασχοληθεί συστηματικά με τον έλεγχο ενσωμάτωσης ή εφαρμογής του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου. Ωστόσο, η γενικότερη τάση, όπως διατυπώθηκε με σειρά ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου κατέστη σαφές ότι δίδεται προτεραιότητα στην αναθεώρηση και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας οδηγεί νομοτελειακά στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει και εμείς ως θεσμός με ελεγκτικέ αρμοδιότητες να δραστηριοποιηθούμε στην αξιολόγηση της εφαρμογής των υποαναθεώρηση νομοθετημάτων. Όπως προανέφερα, η ανταλλαγή καλών πρακτικών θα βοηθήσει ιδιαίτερα εμάς που βρισκόμαστε στο αρχικό αυτό στάδιο προκειμένου να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Παραθέτω εδώ μερικές ιδέες. Αρχικά πιστεύω θα πρέπει να γίνει καταγραφή και μελέτη των περιπτώσεων παραβάσεων που είτε εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή βρίσκονται σε πιο αρχικό στάδιο, ας, πούμε της αιτιολογισμένης γνώμης, έτσι ώστε να αποκτήσουμε σαφή εικόνα των αιτιών της καθυστέρησης ή της πλημελούς εφαρμογής. Είναι λόγοι οικονομικής φύσης, λόγοι διοικητικών δυσλειτουργιών, έλλειψης συντονισμού μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων, αντιδράσεις κοινωνικών ομάδων ή ομάδων συμφερόντων και για να εντοπίσουμε τους τομείς της νομοθεσίας που παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα. Η ελεγκτική μας λειτουργία θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική αν υπήρχε ανάλογη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν δέχεται καταγγελίες πολιτών θα μπορούσε, για παράδειγμα, η καταγγελία που μπορεί να υποβάλει απευθεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε Ευρωπαίος πολίτης να κοινοποιείται ταυτόχρονα και σε μια ειδική για το σκοπό αυτό γραμματοθυρίδα του Κοινοβουλίου. Αντίστοιχα, θα ήταν χρήσιμο, αν υπήρχε επαρκής διοικητική υποδομή, να κατατάσσονται οι αναφορές πολιτών που κατατίθενται στη Βουλή και απευθύνονται προς υπουργού, όχι μόνο με χρονολογική σειρά όπως γίνεται τώρα, αλλά και κατά θέμα, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις που αφορούν προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας. Τέλος, θα βοηθούσε η ακρόαση σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπροσώπων κοινωνικών φορέων ή της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους τόσο για την υφιστάμενη νομοθεσία, όσο και για υποσυζήτηση σχέδια νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ευρύτερη αλληλοενημέρωση. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα μέσα αντίδραση των κοινοβουλίων αναφορικά με ενδεχόμενος παραβιάσεις της αρχής της αναλογικότητας μας αποθαρρύνει πολλές φορές να ασχοληθούμε συστηματικά με μια νομοθετική πρόταση προβληματική ως προς την αναλογικότητα και να εκδώσουμε γνώμη αφού γνωρίζουμε εκ των, προτέρων ότι δεν θα ληφθεί υπόψη. Αυτό έχει δύο αρνητικές συνέπειες. Αφενός, ευνοείται η ταχεία υιοθέτηση νομοθετικών προτάσεων, οι οποίες είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε ορισμένα κράτη-μέλη λόγω δυσανάλογου διοικητικού βάρους ή οικονομικών επιπτώσεων που συνεπάγονται και αφετέρου ο όγκος των προτάσεων που καταλήγουν σε συζήτηση μειώνεται αισθητά αφού περιοριζόμαστε σε όσες παρουσιάζουν προβλήματα με την αρχή της επικουρικότητας, οι οποίες και είναι ελάχιστες. Συμπερασματικά, η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 260 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέτεινε στην επιτάχυνση της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό, αλλά για να επιτευχθεί ορθή και υποφελής εφαρμογή του χρειάζεται πάνω απ' όλα ενημέρωση των πολιτών και οικειοποίηση των προτινόμενων μέτρων. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή των κοινοβουλευτικών, τόσο των εθνικών όσο και των ευρωβουλευτών, στα αρχικά στάδια διαμόρφωσης της νομοθεσίας είναι καθοριστικής σημασίας. Σας ευχαριστώ. Bene. Moltissime grazie, eh, onorevole Chiotis. Ora sono lieta di dare la parola al prossimo ospite, l'onorevole Branner, deputato del Parlamento tedesco. Anche lei dieci minuti di tempo. Grazie. Ο κύριος Μπράντερ από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αγαπητέ ε, κύριε, αγαπητοί κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση να σας παρουσιάσω την ε, σκοπιά της Γερμανικής βουλή. Ονομάζομαι Μπράντνερ, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Προστασίας των Καταναλωτών. Είχα την ε, ευκαιρία να ακούσω τους ε, προλαλήσαντες με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και λοιπόν που ήρθε η δική μου ε, σειρά θα σας ενημερώσω για την περίπτωση της Γερμανίας. Υπάρχει λοιπόν η διαδικασία συναπόφασης, το νομοθετικό έργο μοιράζεται ανάμεσα ε, στο, στην Bundestag, Νομοσπονδιακή Ομοσπονδιακή Βουλή και το Bundestag, το Ομοσπονδιακό ε, ε, Συμβούλιο. Στο άρθρο 23 του Συντάγματος αυτή η συνεργασία είναι θεσμοθετημένη, αλλά αναφέρεται επίσης και ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει υποχρέωση ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη γερμανική Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση της ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο γερμανικό δίκαιο, όμως ε, το αν αυτό συμβαίνει ε, ευχάριστα είναι τελείως ε, διαφορετικό θέμα. Υπάρχει δευτερογενές δίκαιο το οποίο παράγεται και από τα ε, κράτη-μέλη. Επίσης, ε, σε ό,τι φορά τις οδηγίες ε, και τους κανονισμούς, το δευτερογενές δικαίωμα φορά κυρίως τις οδηγίες και όχι τους κανονισμούς. Τα όρια ανάμεσα σε μια οδηγία και σε έναν κανονισμό νομίζω πως έγιναν σαφέστερα τα τελευταία χρόνια. Από τη μία υπάρχουν σαφείς διατάξεις για το τι συνιστά μια οδηγία και από την άλλη υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κανονισμοί που έχουν πάρα πολλές ε, πάρα πολλές ε, διατάξεις. Οπότε λοιπόν δεν είναι και τόσο σαφή τα όρια. Όμως ο Ευρωπαίος νομοθέτης έχει λοιπόν οδηγίες και κανονισμούς στους οποίους πρέπει να ενσωματώσει ε, η γερμανική κυβέρνηση. Καταρχάς η νομοθετική ε, ρυθμιστική αρμοδιότητα προκύπτει από το γερμανικό σύνταγμα. Η νομοθετική αρμοδιότητα ανήκει στην Ομοσπονδία λοιπόν. Ακριβώς σε μια που το νομοθετικό έργο αφορά την ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Επίσης υπάρχουν τα τοπικά κοινοβούλια, τα οποία επίσης ε, ασκούν ενεργά νομοθετικό έργο, όπως για παράδειγμα το, το κοινοβούλιο της ε, Θουρυγγίας, στο Πιανίκο. Υπάρχουν λοιπόν επικαλύψεις ε, στο νομοθετικό έργο και η Ομοσπονδία σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να τις ε, ενσωματώνει στην ολότητά τους. Οι διάφορες ελλείψεις που εντοπίζονται στην ε, γερμανική νομοθεσία αντιμετωπίζονται μέσω, μιας, μέσω ειδικής νομοθεσίας και μέσω μιας ειδικής επιτροπής. Έπειτα, Το ερώτημα μένει, ε, ε, παραμένει για το εάν μια οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται α, ε, και να ψηφίσετε από το Κοινοβούλιο ή από την κυβέρνηση. Υπάρχουν δύο στάδια ενσωματώσεις μιας οδηγίας ή ενός κανονισμού. Αυτό καταρχάς ενσωματώνεται μια οδηγία, ένας κανονισμός μόνο εφόσον εγκριθεί και υπερψηφιστεί από την Βουλή. Οι κανονισμοί απαιτούν, ε, δηλαδή, για τους κανονισμούς δηλαδή απαιτείται ένα σαφές ε, νομικό πλαίσιο. Η νομοθετική διαδικασία είναι η συνήθις νομοθετική διαδικασία που συμβαίνει όταν ψηφίζεται και ένας εθνικός νόμος. Το ίδιο γίνεται και, στο, και στην περίπτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τώρα νομίζω ότι η επιλογή του νομικού μέσου είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, δηλαδή ε, οδηγία ή κανονισμός. Νομίζω πως στις Βρυξέλλες παρατηρείται μία τάση ε, ότι η Επιτροπή κατά, τη διάρκεια, την διάρκεια της άσκησης του δικαιώματος πρωτοβουλίας ε, προτιμά τον κανονισμό και λιγότερο οδηγία. Ε, αυτό μας δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία της ε, EURLEX από το 2017, ε, τα οποία έχουν αναλύσει τις νομικές πράξεις της νομοθετικής διαδικασίας και βλέπουν ότι οι κανονισμοί υπερτερούν των οδηγιών κατά έξι φορές. Έξι φορές περισσότεροι κανονισμοί από ότι οδηγίες. Αυτά σε ό,τι φορά τη νομική βάση. Και ε, το ίδιο παρατηρήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την επιλογή λοιπόν να επιλέξει ανάμεσα σε μια οδηγία και έναν ε, κανονισμό. Η βάση για την επιλογή της αποτελεί η αρχή της αναλογικότητας. Το άρθρο 296 αναφέρεται στις ε, περιπτώσεις ε, όπου τα όργανα θα, όπως είπε και ο ε, προγραλής σας, θα αποφασίσουν για το νομικό μέσο που θα χρησιμοποιήσουν. Επίσης αναφέρονται και ο τρόπος με τον οποίο θα επιτύχουν τον επιθυμητό ε, στόχο. Προστατεύεται η αρχή της ε, αναλογικότητας. Το θέμα όμως είναι τι ακολουθεί από αυτό το μέτρο. Νομίζω πως ε, σε γενικές γραμμές υπάρχει μία προτίμηση από τα κράτη-μέλη στις από την Κομισιόν στους κανονισμούς. σε γενικές γραμμές ε, βλέπουμε ότι οι οδηγίες θα έπρεπε να είναι το προτιμόμενο ε, μέσο παρά ο κανονισμός αν θέλει να γίνεται σεβαστή απόλυτα η αρχή της αναλογικότητας. διότι λαμβάνουν υπόψη και τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Ακριβώς ό,τι δηλαδή συμβαίνει και με την αρχή της ε, επικουρικότητας. σε πολλές περιοχές η νομοθεσία, σε πολλές περιοχές, από πολλά όμως τα κρατήδια, η νομοθεσία είναι πάρα πολύ παλιά. Πολλές φορές έχουμε νομοθεσία από το 1896, άλλες φορές από τις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει λοιπόν ε, ανάγκη να προσαρμόσουμε ε, την νομοθεσία και γι' αυτό το σκοπό μια οδηγία είναι προτιμότερη από έναν κανονισμό διότι μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ε, ιδιαιτερότητες της δικής μου χώρας. Με Έπειτα υπάρχουν περιπτώσεις ε, νομικής αβεβαιότητας που οδηγούν σε διαδικασίες επιπαραβάση ακριβώ για αυτόν τον σκοπό. Επίσης, πολλές φορές ε, υπονομεύεται ε, ο δίκαιος ανταγωνισμός. Γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχουν ελλείμματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Υπάρχουν ε, αυτές οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά τον εθνικό έλεγχο και η προτίμηση σε κανονισμούς νομίζω πως μπορεί να υπονομεύσει την ίδια την δυνατότητα εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν δηλαδή δυσκολίες τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν έναν κανονισμό ε, περισσότερες από ότι μια οδηγία. Επίσης, νομίζω πως ε, φαίνεται ότι στην ε, νομοθετική ε, διαδικασία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η εφαρμογή, όπως είδαμε όλη τη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο νομίζω πως έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπράνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σεβαστήκατε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Περνάμε τώρα στη συζήτηση. Να ακούσουμε τα σχόλια των βουλευτών. Έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Πρέγω, Βίλαντ. Βίλαντ, παρακαλώ να έχω μια ερώτηση. Να... Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών». Και έχουμε λοιπόν την δυνατότητα της, ε, της προδικαστικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορές ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όταν ε, τα συμβαλόμενα μέρη, για παράδειγμα, ζητούν ε, να, να γίνει προσφυγή στο δικαστήριο. Επίσης, τα ένδικα μέσα διαφέρουν από κράτος σε κράτος, καθώς και η ερμηνεία των ε, νόμων. Ίσως λοιπόν ε, θα μπορούσαν συνάδελφοι να μας δώσουν, δώσουν τις εμπειρίες τους από τη δική τους χώρα. Ευχαριστώ κύριε Κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Αν ο κύριος Δόρμαντ ή η κυρία Σμίθ θέλουν να προσθέσουν κάτι σε σχέση με αυτά που είπαν οι εθνικοί εκπρόσωποι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ο κύριος Μπουσουτήλ ζήτησε το λόγο, τον παρέβλεψα προηγουμένως. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που μας έκαναν τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Όπως είπε και ο προλαλής σας, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να φέρει στο επίκεντρο τον Ευρωπαίο πολίτη. Για τη τελική ανάλυση, όταν δεν εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο, ο χαμένος είναι ο πολίτης. Αυτός βγαίνει χαμένος. Και πραγματικά έχω χάσει τον αριθμό των ε, ψηφοφόρων που έρχονται και με βρίσκουν και που νιώθουν τέτοια απογοήτευση και τέτοιο εκνευρισμό για την πολύ χρονοβόρα διαδικασία προκειμένου να απολαύσουν τα δικαιώματα που τους κατοχυρώνει το ενωσιακό δίκαιο. Και είναι ακόμη πιο ενοχλητικό και απογοητευτικό όταν ε, η αντίσταση προέρχεται από τις αρμόδιες αρχές. Από το ίδιο το δημόσιο που δεν ε, ικανοποιεί, δεν εφαρμόζει τα δικαιώματα των πολιτών. Θα πρότεινα λοιπόν εμείς ως κοινοβουλευτικοί να επικεντρωθούμε περισσότερο στο τι συμβαίνει, το, τι θα έπρεπε να συμβεί στις περιπτώσεις που το ενωσιακό δίκαιο δεν εφαρμόζεται επειδή προσκρούει στην αντίσταση των κυβερνήσεων ή των ε, αρμόδιων εθνικών αρχών. Απέναντι σε μια τέτοια δυσκολία θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. Καταρχήν, ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα στο συνθηκό θα πρέπει να μεριμνά ώστε να εφαρμόζεται σωστά το ενωσιακό δίκαιο. Σε μερικέ περιπτώσεις όμως είναι τεράστια η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τη διαδικασία παραβάσει για την εφαρμογή ε, του ενωσιακού δικαίου. Για παράδειγμα, στην, Επιτροπή, στην ε, πολιτική ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τεράστιε αξιοπιστία ε, και αντιμετωπίζεται ω πραγματικά αμερόληπτο φορέα, αμερόληπτο και έντονο διαμεσολαβητή που εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Σε άλλε περιπτώσει όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται πιο πολιτικοποιημένη και αργοπορεί, κολυσιεργή σε ό,τι αφορά την απέτηση εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη-μέλη. Και μερικέ φορέ οι διαπραγματεύσει γίνονται κάπω παρασκηνιακά, εγκρυπτό και παραβίστο και κάπω αδιαφανώ μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, κρατών μέλων πριν κινήσουν διαδικασίε επί παραβάση. Και δεν είμαι σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκπροσωπεί πάντα το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη και το κοινό αγαθό. Εγώ θα ήθελα να είναι όντω και πλήρως αμερόληπτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα ζητήματα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και για την εκκίνηση διαδικασιών επί παραβάση. Αυτή θα είναι η Επιτροπή που γνωρίζουμε στην ε, πολιτική ανταγωνισμού και θα θέλαμε να είναι σε όλες τις πολιτικές έτσι, αμερόληπτη θεματοφύλακα των συνθήκων. Επίσης, συμφωνώ με τα σχόλια που έκανε η Διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας ε, που, αν κατάλαβα καλά, πρότεινε το πρωί ένα είδος διευρυμένης συνεργασίας μέσω κάποιου θεσμοθετημένη δομή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Τέτοιου είδου συνεργασία θα ήταν σημαντική για να ενισχυθεί η θέση του Ευρωπαίου πολίτη, κυρίως όταν α, αντιμετωπίζει την αντίσταση των εθνικών αρχών και μερικές φορές νιώθει ανήμπορος ο πολίτης και δεν μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Ίσως λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών και η Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να εγκρίνουν το, τη σύσταση της εκπροσώπου της νομικής υπηρεσίας και να θεσμοθετηθεί ένα, ένα είδος συνεργασίας με κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, ώστε οι κοινοβουλευτικοί και των 28 χωρών να συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εφαρμόζεται σωστά το ενωσιακό δίκαιο, ειδικά στις περιπτώσεις που έχουμε αντίσταση των εθνικών αρχών για αυτή την εφαρμογή. Σας ευχαριστώ πολύ Υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις από πλευράς των παρεμπιστημένων. Κυρία Ρωσίνη, παρακαλώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους φτάνει κανείς στην ε, παράβαση Μπορώ να πω ότι το Εθνικό Κοινοβούλιο βιώνεται από τους πολίτες ως τόπος εκπροσώπησης. Πολύ συχνά, συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αδίκως συχνά βιώνεται από τους πολίτες σαν κάτι επιβεβλημένο, σαν μια επιβολή. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί το Ιταλικό Κοινοβούλιο βρίσκεται ανάμεσα στις πληγάδες των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτή είναι μια πραγματική κατάσταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο καθηγητής Γκέστα. Θα πρέπει να καταφέρουμε να προηγηθούμε των καιρών μας. Θα πρέπει να καταφέρουμε τα Ευρωπαϊκή Κοινοβούλια πριν να λάβουν τις προτάσεις, να έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν ε, ε, ε, να μπορούν να εκφράσουν τους πολίτες τις, τις τοπικές κοινότητες πάρα πολλές φορές ε, ε, πολλοί ζουν καθ' υπερβολή την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν προβλήματα. Η Ευρώπη είναι φτιαγμένη και από μικρές πραγματικότητες και θα πρέπει να τις προφυλάξουμε προκειμένου να κρατήσουμε άρρηκτα δεμένο ε, δεμένες της κοινότητας, αυτή, Αυτή είναι μια εντολή που έχουμε και είναι κάτι που νιώθω βαθιά. Πιστεύω ότι το να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ανιούσα φάση, τη φάση των προτάσεων μεταξύ των άλλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να αποφύγει το να ξεσπάσουν συγκρούσει μεταξύ των τριών αυτών επιπέδων πολιτών, Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Και η τελευταία πρόταση, που, η οποία με βρίσκει σύμφωνο, όπως και άλλους ε, βουλευτές, αφορά τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων ενδεχομένως ε, δεν έχει εξελιχθεί πλήρως ε, αυτό. Αυτό θα πρέπει να έχει στόχο να διευκολύνουμε οι οδηγίες και οι κανονισμοί ακόμα περισσότερο που εφαρμόζονται άμεσα να μην βιώνονται σαν κάτι επιβεβλημένο εκ των άνωθεν. Υπάρχει ανάγκη από τους ίδιους τους πολίτες να ακούσουν περισσότερο ε, να ακουστεί περισσότερο φωνή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεσμεύομαι να αναζητήσω μια βελτίωση αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρωσίνη. Έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο καθηγητές, αν θέλουν σε δύο, δυόμιση λεπτά, πολύ λακωνικά να κάνουν σύντομα σχόλια ε, σχετικά με ό,τι υπόθηκε από τους εθνικούς βουλευτές. Ο καθηγητής Βέρμα, παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις σας. Αν κατάλαβα καλά την απορία του κυρίου Βίλαντ εδώ θα έπρεπε να συζητούμε την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, όχι μόνο την ενδυνάμωση των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και το πώς οι πολίτες ε, ε, μπορούν να βρουν το δρόμο τους στις διάφορες διαδικασίες. Να προσφύγουν στο δικαστήριο, για παράδειγμα, ζητώντας ε, θέση προδικαστικού ερωτήματος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα, γιατί αυτό που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στις κατοχώρες φυσικά, είναι ότι τα δικαστήρια και οι δικαστές ε, είναι διστακτικοί απέναντι στη χρήση του προδικαστικού ερωτήματος, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, παρόλο που είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες να τίθενται τέτοια προδικαστικά ερωτήματα από τα δικαστήρια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πολύ συχνά οι διάδικοι σε διάφορες δίκες στην Ολλανδία ζητούν να τεθεί προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί θέλουν να ξέρουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου για το θέμα τους. Και μερικές φορές το αίτημά τους δεν γίνεται δεκτό. Δεν παραπέμπεται το προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τον Εθνικό Δικαστή, γιατί ο εθνικό Δικαστής νομίζω ότι ξέρει τη σωστή ερμηνεία. Προσοχή λοιπόν, ίσως θα πρέπει πιο σωστά, πιο συχνά να τίθεται τέτοια προδικαστικά ερωτήματα για να διευκρινίζεται η ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου. Οπότε εκεί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πολύ εύστοχο το ερώτημα του κύριου Βίλαντ. Επίσης, ο κύριος Μπουσουτήλ και η κυρία Ρωσίνη έθεσαν κάποιες ερωτήσεις. Εγώ έχω ένα σχόλιο εδώ, γιατί είναι θέμα που αφορά περισσότερο την κυρία Σμιθ τις δικές της αρμοδιότητες και γνώσεις. Μία έρευνα που έγινε στην Ευρώπη για το πώς τα κράτη-μέλη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο ε, τις κοινοτικές οδηγίες. Ε, ε, θα σας πω κάτι που γνωρίζω χωρίς να κατανομάσω την χώρα. Πήγαμε σε μία χώρα και συζητούσαμε με έναν αρμόδιο και όπως είπε ο Έλληνας εκπρόσωπος, ε, είστε στην ενδέκατη θέση του πίνακα επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την μεταφορά. Και τότε ένας υψηλόβαθμος ε, αξιωματούχος ε, από τη Γενική Διεύθυνση είπε «Κοίτα, ε, δείξτε το μου, αποδείξε το μου». Ενδέκατη θέση αποκλείεται, σίγουρα είμαστε καλύτεροι. Βλέπετε το στοιχείο της ε, Realpolitik εδώ. Στρατηγικός τους ε, στόχος είναι να είναι καλοί μαθητές και να μεταφέρουν αμέσως τις οδηγίες ε, στο εθνικό δίκαιο. Αλλά μερικές φορές αυτό έχει και μια αρνητική πλευρά. Αν δεν το κάνουν όλοι αυτό και αν δεν όλοι μεταφέρουν τις οδηγίες, τότε μπορεί να δημιουργούνται συνθήκες αθέμη ανταγωνισμού και να πλήττονται οι ε, επιχειρήσεις. Θα πρέπει όλοι να ε, πασχίζουν για άμεση μεταφορά. Δεν αρκεί μία πανηγυρική δέσμευση ή υπόσχεση. Γιατί σίγουρα αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας ε, είναι κάτι καλό, αλλά ίσως χρειάζεται κάτι περισσότερο. Περισσότεροι κανονισμοί αντί για Δεν έχω πιστεί από τον ε, εκπρόσωπο της Γερμανίας, τον κοινοβουλευτικό της Γερμανίας, που είπε ότι ε, είναι κακή ιδέα να έχουμε περισσότερους κανονισμού από ό,τι οδηγίε. Διαφώνω, μερικέ φορέ βοηθάνε οι κανονισμοί. Πάντω κάτι θα πρέπει να κάνουμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία της μεταφοράς των κοινοτικών οδηγιών. Γιατί εδώ μερικές φορές, παίζονται και στρατηγικά παιχνίδια. Κυρία Σμίτ, ε, έχουμε ένα λεπτό, ένα λεπτό γρήγορα σας παρακαλώ. Καλώς. Ε, πολύ σύντομα για τα προδικαστικά ερωτήματα. Όντως αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Τα προδικαστικά ζητήματα σπάνια είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιβεβαιώσει ε, το και να κατοχυρώσει τα δικαιώματα πολίτη. Γιατί είναι χρονοβόρε, δαπανηρέ διαδικασίε, απρόβλεπτη έκβαση, γιατί και εδώ είναι θέμα διακριτική ευχαίρεια του δικαστού. Οπότε δεν είμαι σίγουρη για το πόσο ε, θετικά είναι τα προδικαστικά ερωτήματα. Ούτω ή άλλω πολλές φορές ε, στηριζόμαστε στη διπλή διαδικασία των επιβαραβάσεων διαδικασιών και των προδικαστικών ερωτημάτων, αλλά μερικές φορές και αυτό το διτό σύστημα είναι ανεπαρκές. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αμεροληψίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, έχω γράψει και βιβλίο επικρίνοντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μεροληπτική τη μερικέ φορέ τάση. Αλλά τώρα θα την υποστηρίξω γιατί η Ευρωπαϊκή Πολιτική είναι πολιτικό σώμα με πολιτικέ προτεραιότητε. Οπότε λογικό είναι να εκείνη η διαδικασία σε επιβαραβάσει ανάλογα με τι πολιτικέ προτεραιότητε. Γιατί οι πόροι τη είναι περιορισμένοι και δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Οπότε θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Γιατί τώρα φαίνεται αμερόληπτη στο δίκαιο ανταγωνισμού. Γιατί εκεί είναι ένα ανεξάρτητο διαιτητή ανάμεσα σε δύο εμπορικέ ε, σε δύο εμπορικού αντιπάλους. Και εδώ είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα, η κατάσταση στον ανταγωνισμό. έξω και η αμεροληψία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά και βάζω τελεία εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω και στο μέλλον να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να ξαναμιλήσουμε για αυτά τα θέματα, επειδή βρισκόμαστε ενώπιον προκλήσεων για τη νέα νομοθετική περίοδο. Ε, ειλικρινά λυπάμαι, δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. number. Okay, thank you very much. Thanks. So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι που συζητάτε μεταξύ, μας, μεταξύ σας κάτι που δείχνει πόσο χρήσιμες είναι τέτοιου είδους συνεδριάσεις και συναντήσεις. Δυστυχώς όμως μας πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε, να περάσουμε στο τρίτο πάνελ που έχει τίτλο «Το ρόλο των καταγγελιών των προσφυγών προς το διαμεσολαβητή, το συνήγορο του πολίτη και αναφορές στα κοινοβούλια ως μέσα εντοπισμού παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, την κυρία Έμιλη Οράιλη, για να μας κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι κοντά σας για αυτό το πάνελ που φυσικά μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο ρόλος ε, του Διαμεσολαβητή και τη Επιτροπή Αναφορών για τον εντοπισμό παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου. Όπως ξέρετε, ο Διαμεσολαβητής βρίσκεται μεταξύ των πολιτών και της διοίκηση και η θέση του μας επιτρέπει να βρίσκουμε ακριβώς που αναδύονται προβλήματα. Και γι' αυτό με συστάσει και άλλους τρόπους προσπαθούμε να έχουμε μια πιο διαφανή και υπόλογη δημόσια υπηρεσία. Φυσικά θέλουμε να χρησιμοποιούμε την ήπια δύναμη, το soft power και χάρη στην έρευνα και τον έλεγχο που κάνουμε εντοπίζουμε τα προβλήματα και με την επιρροή μας προσπαθούμε να επιφέρουμε αλλαγέ. Μερικές φορές με μια καταγγελία μπορεί να εντοπιστεί ένα πρόβλημα που επηρεάζει μια ευρύτερη ομάδα οι παρόμοια, θέμα, παρόμοια καταγγελίες μπορούν να επισημαίνουν ένα συστημικό πρόβλημα. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποίησα τη δυνατότητα πρωτοβουλίας που έχω για να ξεκινήσω ευρύτερες στρατηγικές έρευνες και να εξετάσω συστημικά ζητήματα από το να έχω ξεχωριστέ έρευνε για κάθε καταγγελία ξεχωριστά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που νομίζω ότι αγγίζει την καρδιά του σημερινού θέματο είναι η στρατηγική μου έρευνα για το πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει καταγγελίε επί παραβάση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ε, Προγράμματο EU Pilot που στόχο έχει να εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο παραβίαση ενωσιακού δικαίου για να αποφευχθεί προσφυγή σε διαδικασίε επιπεραβάση. Μετά όμω από πολλέ καταγγελίε που έγιναν για το σχέδιο Pilot, προσπάθησα να υιοθετήσω μια πιο οριζόντια στρατηγική. Η στρατηγική μου έρευνα κάλυψε πολλά προβλήματα. Καταρχήν ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τη διαδικασία ε, εξέταση των καταγγελιών και επίση ε, έκανε κάποιε συστάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει τη σχέση τη με του καταγγέλλοντε και να ενισχύσει τη διαφάνειά τη. και διαπίστωσα ότι πολλά προβλήματα προέκυψαν από την έλλειψη κατανόηση για την επεξεργασία των καταγγελιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αποτυχία μερικέ φορέ Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί στι προσδοκίε των πολιτών ενώ ε, προσπαθεί πραγματικά να διορθώσει ένα διαδικαστικό πρόβλημα. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακόπτει ή δεν εκείνη μια διαδικασία, θα πρέπει να εξηγείται όντω στον καταγγέλλοντα γιατί δεν το έκανε. Η δεμή ε, εκνευρίζει και απογοητεύει τους καταγγέλλοντος. Για παράδειγμα, είχαμε μια καταγγελία για την εφαρμογή από τη Γερμανία τη οδηγία για την ιδιωτικότητα. Οπότε σύστησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε να δικαιολογήσει επαρκώ γιατί δεν έκανε την ε, επεξεργασία, είτε να την ξανανοίξει. Τελικά δόθηκε μια εξήγηση, αλλά όχι πλήρω αιτιολογημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι άλλο ε, που βοηθάει στην ανείχνευση παραβιάσεων είναι η ε, άρνηση πρόσβασης ε, σε δημόσια έγγραφα. Συνήθως αυτοί που ζητούν πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα είναι γιατί θέλουν να πιστήσουν την προσοχή μας σε κάποιο πρόβλημα. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι πρόσφατη καταγγελία ενός ευρωβουλευτή που ζητούσε πρόσβαση στα πρακτικά συνεδριάσεων της Ρυθμιστικής Επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές των οχημάτων και ήθελε ε, να ε, έχει πρόσβαση στις εκθέσεις στα πλαίσια της έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο Dieselgate. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα να δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτά τα πρακτικά και κυρίως στις θέσει των εκπροσώπων των κρατών μελών. Όπω είπα και το πρωί, οι πολίτε θα πρέπει να έχουν δικαίωμα για το τι κάνουν οι κυβερνήσει του και όταν βρίσκονται στι Βρυξέλλε. Και μάλιστα μέσω του δικτύου ε, διαμεσολαβητών δίνουμε μία άλλη δίωδο για να αντιμετωπιστούν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου γιατί από το δίκτυο μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες σε μένα για ευρωπαϊκά θέματα που εντοπίζονται στα πλαίσια των ερευνών των συνηγόρων του πολίτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρκετά συνεργάσιμη σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες αυτές. Έτσι μπορούμε να διευκολύνουμε εθνικές και περιφερειακές έρευνες που οι δεμοί δεν θα γίνονταν εύκολα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ήταν μια έρευνα του Ομοσπονδιακού ε, Βελγίου Συνηγόρου του Πολίτη για την οδηγία και την οικογενειακή επανένωση. Και μάλιστα δεν ήμουν ε, στην Ιρλανδία συνηγόρος του πολίτη, ε, είχα θέσει ζητήματα ε, γεωργικών ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επίσης έχουμε πολλές φορές παράλληλες πρωτοβουλίες και έρευνες μαζί με τους συναδέλφους του δικτύου διαμεσολαβητών για να δούμε κάποια θέματα στα οποία μπλέκονται περιφερειακές ή ε, εθνικές αρχές. Για το πώς, για παράδειγμα, οι Ευρωπαϊκοί πώς αντιμετωπίζονται και εφαρμόζονται οδηγίες για δραστικές ουσίες που ε, μειώνουν το όζο στην ατμόσφαιρα. Επίσης, σε θέματα εξαγωγικών επιστροφών και κάποιες καταγγελίες που έγιναν για, για τις υποχρεώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς α, ε, α, ε, μερικοί ετούντες άσυλο που απορρίθηκε η, το αίτημά τους επιστρέφουν στη χώρα τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις επισήμανα παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου. Και έχω και άλλα παραδείγματα από το έργο περιφερειακών ή εθνικών συνηγόρων του πολίτη στα πλαίσια των ε, αναφορών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αναφορών. Σας ευχαριστώ κυρία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, διακεκριμένοι συνάδελφοι από την Επιτροπή Αναφορών, θα δούμε τώρα πώς βλέπουμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η Επιτροπή Αναφορών κάθε χρόνο ετοιμάζει μια γνωμοδότηση που αφορά την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού δικαίου και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα και με μερικούς συναδέλφους από άλλες επιτροπές έχουμε θαυμάσια συνεργασία με το γραφείο της ε, Διαμεσολαβρήτριας και βεβαίω έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Γι' αυτό το λόγο οργανώσαμε αυτή την συνάντηση για να έχουμε μια συνάντηση με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και με τους διαμεσολαβητές. Βεβαίως επιθυμία μας είναι να συνεχιστούν αυτές οι δραστηριότητες από το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή ήταν μία σύντομη δήλωση από την Επιτροπή Μεταφορών. Τώρα θα ήθελα να παρατηρήσω τον ε, πραγματογνώμονα από το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, τον κύριο ε, Ταβιάγο Τιμπούρσιο, για να μιλήσει για το ρόλο του διαμεσολαβητή. Κύριε Τιμπούρσιο, ο λόγος ανήκει σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είναι τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσω για ένα τόσο ευγενές θέμα, για το ρόλο των διαμεσολαβητών σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των, παραβιάσεων, των παραβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, παρουσίασή μου, στην παρουσίασή μου θα ακολουθήσω τις ε, διαφάνειες που έδειξα και που αφορούν τις ε, διαφορές μεταξύ των καταγγελιών και των ε, αιτήσεων. Μετά θα παρουσιάσω μερικές βέλτιστες πρακτικές και θα κάνω και συστάσεις. Σε ό,τι αφορά τις ε, καταγγελίες και τις αναφορές, θα ήθελα να παραθέσω δύο τρόπους που έχει στη διάθεσή του ο ε, ο πολίτης προκειμένου ε, να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να οριοθετηθεί το πλαίσιο αυτών των δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε σκοπό να δώσουμε φωνή στους πολίτες αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το θέμα είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία, όχι να ληφθεί μια απόφαση. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει μία γνωμοδότηση, αλλά στην πραγματικότητα τα δικαστήρια είναι εκείνα που αποφασίζουν στην περίπτωση των δικαστηρίων. Η διαδικασία είναι πιο διακριτική Ακόμα και αν υπάρχουν οι ειδικοί που αναφέρονται στη τελική δήλωση του διαμεσολαβητή. Πρόκειται για παράλληλα δικαιώματα, δίδυμα δικαιώματα, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Υπάρχει ένα ε, δίκαιο ε, συμβατική συμμετοχής η δέσμευση που απαιτείται σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται. Θα πρέπει γραπτός να υποβάλλεται η καταγγελία και στην περίπτωση του διαμεσολαβητή μπορεί η καταγγελία να είναι και προφορική. Και τα άλλα δικαιώματα, το δικαίωμα ψήφου, είναι αποκλειστικό δικαίωμα του πολίτη και αυτό είναι σημαντική στιγμή για τα θεσμικά όργανα. Και ε, εδώ η συχνότητα είναι περιορισμένη που να εναπόκειται το δικαίωμα αποκλειστικά μόνο του πολίτη, στον πολίτη. Πολλές φορές εναπόκειται στα θεσμικά όργανα. Αλλά γι' αυτό σε μερικές περιπτώσεις ε, ζητούμε την αιγίδα ή την ε, διαμεσολάβηση του διαμεσολαβητή. Και σίγουρα ο καταγγέλων ή ο αναφερόμενος ζητά μία απάντηση, μία, ένα feedback στις επαφές που έχει με τα θεσμικά όργανα, γράφοντας επιστολές για παράδειγμα. Και ε, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Έχουμε την άμεση δημοκρατία και την αμεγώς αντιπροσωπευτική δημοκρατία ή την υπερασπιστική δημοκρατία που δίνει ευκαιρία συμμετοχής στους πολίτες, αλλά στη τελική ανάλυση την απόφαση τη λαμβάνουν οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, ξεκινούμε με μία ανησυχία που σχετίζεται ιστορικά με το θέμα αυτό. Καταρχήν το θέμα της συμπερίληψης. Μερικές φορές έχουμε ομάδες που δεν ακούγεται η φωνή τους και ε, στην πράξη δεν ε, έχουμε πάντα αυτή την ε, πολυμορφία. Για παράδειγμα, κάποιοι συγγραφείς μιλούν για τις αδυναμίες αυτής της υπερασπιστικής δημοκρατίας, γιατί μερικές φορές χρησιμοποιούνται από εκείνους που έχουν την περισσότερη ισχύ και αυτοί ασκούν υπέρμετρα αυτό το δικαίωμα. Ε, Επίση, δεν έχουμε ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε, στα διάφορα θεσμικά όργανα. Φαίνεται και εδώ η διαφορά στα δύο φύλλα. Βέβαια, το σύστημα των αναφορών έχει ξεχρονιστεί την τελευταία δεκαετία και δείχνει ότι υπάρχει σημαντική υπερεκπροσώπηση των ανδρών. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να είναι πιο πολύμορφη. Ε, για παράδειγμα, ο συνήγορος του πολίτη της Λιθουανίας ε, κάνει έρευνα του πληθυσμού κάθε χρόνο και με τις ε, πληροφορίες που συγκεντρώνει μπορεί να διοργανώσει εκστρατείες προς ομάδες που δεν γνωρίζουν και πολύ καλά το ρόλο του συνήγορου του πολίτη. Επίσης ε, και στη Βόρεια Ιρλανδία ε, ο διαμεσολαβητής ε, εκπονεί την έκθεση της ισότητας ανάλογα με τις διαφορές φύλων, εθνοτικής καταγωγής, πολιτικών απόψεων και ούτω καθεξής. Και σίγουρα ε, φαίνεται ότι δεν είναι γενικευμένη η προσφυγή στο, δίκαιο της, στο δικαίωμα της αναφοράς ή στο δικαίωμα της καταγγελίας και μερικές φορές δεν χρησιμοποιούν επαρκώς οι πολίτες ε, αυτά τα μέσα. Γι' αυτό τέτοιου είδους εκθέσεις, αν αυτές που κάνουν οι συνήγοροι του πολίτη, είναι χρήσιμες για να εντοπιστούν ε, οι αδυναμίες και να προταθούν κάποιες βελτιώσεις. Τώρα, η σημασία της διαδικασίας της υποβολής αναφορών ε, φαίνεται στις διάφορες πρακτικές, κυρίως με τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες, μέσα των ακροάσεων και καθορίζοντας ε, την βέλη των συζητήσεων με συμμετοχή ε, βουλευτών, προσώπων της κυβέρνησης ή υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων. Και μάλιστα έχουν σημαντικό αντίκτυπο όταν μεταδίδονται είτε στο διαδίκτυο είτε να μεταδίδονται στην τηλεόραση. Αυτό συμβαίνει με τις συνεδριάσεις Τη Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Πορτογαλία. Η αναμετάδοση στο κανάλι της Βουλής της Πορτογαλίας. Επίσης, στην Ουαλία ε, φάνηκε το, η επιθυμία των Ουαλών πολιτών να έχουν μια πιο προσωπική επαφή στη διάρκεια της εξέτασης των αναφορών. Επίσης, έχουμε διάφορα κατόφλια εδώ σε ό,τι αφορά την δημοσίευση ή την δημοσιότητα που λαμβάνουν στη τέτοιου είδους συζητήσεις. 4.500 υπογραφές απαιτούνται στο Λουξεμβούργο, 1.000 υπογραφές στο, στην Πορτογαλία, 50.000 απαιτούνται στη Γερμανία. Βέβαια, όταν έχουμε τέτοια κατόφλια, υπάρχουν και κάποια κίνδυνοι. Μερικέ φορέ αυτά τα κατόφλια δημιουργούν πρόσκομα στην πρόσβαση των πολιτών σε τέτοιε δυνατότητε και είναι άνηση ε, η συμμετοχή, η, η έκταση που δίνεται ανάλογα με το ο καταγγέλων είναι από την Ήπεθρο ή από ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Επίσης, το πόσο ρεαλιστικό είναι το αίτημα. Βέβαια υπάρχουν και κάποια πλεονεκτήματα. Από τη στιγμή που φτάσουμε σε αυτό το κατόφλι, ο πολίτης έχει πρόσβαση σε, αυτά, σε αυτούς τους μηχανισμούς, στην ακρόαση, στη συζήτηση, στην δημόσια αναμετάδοση και γίνεται ένα είδος ε, ε κοινή εξέτασης. Σε ό,τι αφορά τα κατόφλια και η συνήγοροι του πολίτη και οι επιτροπέ αναφορών λαμβάνουν πολλέ φορέ συλλογικέ καταγγελίε ή αναφορέ. Έτσι, εμ, διευρύνεται η ομάδα των πολιτών με τις οποίες έχουν, έχουν επαφές. Επίσης έχουμε κάποιες επίσημες επιγραμμικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν τις ε, υπογραφές. Και έτσι οι συντάκτες των ε, αναφορών ή των καταγγελιών ε, μοιράζονται το πρόβλημά τους με ένα ολόκληρο στερέωμα υπογραφών Επίσης, οι ηλεκτρονικές αναφορές είναι σημαντικό λιθαράκι στη σχέση μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων. Και έτσι, χάρη στις ηλεκτρονικές ε, αναφορές, φτάνουμε σε πολίτες που μέχρι στιγμής δεν είχαν μεγάλη εκπροσώπηση, νέους ή πιο περιθωριοποιημένους. Βέβαια, η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες είναι άνηση, και εδώ λοιπόν μπορούμε να έχουμε υπερεκπροσώπηση κάποιων τμήματων πληθυσμού ε, λόγω αυτού του ψηφιακού χάσματος που υπάρχει. Γι' αυτό και θα πρέπει να διασφαλίσουμε παραδοσιακές μορφές συμμετοχής όπως είναι οι έγγραφες αναφορές ή τηλεφωνικές καταγγελίες. Έτσι θα περιορίσουμε την ανισότητα λόγω ψηφιακού χάσματος. Επίσης ε, αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα ε, με μετέτρεψαν μια διαδικασία που ήταν προσωπική σε μια δημόσια διαδικασία, γιατί δίνουν πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ε, για την πορεία μιας αναφοράς ή μιας καταγγελίας, για τις ερωτήσεις που υποβάλλονται στην κυβέρνηση, για τις απαντήσεις που δίνει η κυβέρνηση, οι δημόσιες αρχές και το καθεξής. Επίσης, ε, ε, έχουμε ένα μέσο επικοινωνίας με την κοινωνία που δεν υπήρχε προηγουμένως. Και αυτό είναι μεγάλο κίνητρο για την βελτίωση των διαδικασιών αυτών. Ε, ένα μέσο που χρησιμεύσε για την διεύρυνση αυτών των μέσων είναι τα μέσα κοινωνική ε, δικτύωση, γιατί δίνουν πληροφορίε για το έργο των θεσμικών οργάνων και ε, επιτρέπουν το σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο του έργου των συνηγόρων του πολίτη. Μέσω του Twitter, για παράδειγμα, παρόλο που σπάνια χρησιμοποιούνται αυτέ οι ε, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης από, τις, από τους συνηγόρους του πολίτη, με μερικές εξαιρέσεις. Ε, αντίθετα, χρησιμοποιείται από τις Επιτροπές Αναφορών, γιατί είναι ένας καλός τρόπος ε, διαχείρισης των πληροφοριών. Βέβαια, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται μονόδρομα εδώ θα μπορούσαμε να προωθήσουμε ένα καλύτερο διάλογο, πραγματικό διάλογο με τους πολίτες, ε, μεταξύ πολιτών δηλαδή και επιτροπών αναφορών ή συνηγόρων των πολίτη, χάρη σε αυτές τις πλατφόρμες. Ε, ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών για, τη, για το ρόλο αυτών των θεσμικών οργάνων, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Η επικοινωνία εδώ έχει κέριο ρόλο. Μία επικοινωνία που δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην μετάδοση κάποιων πληροφοριών, αλλά θα πρέπει να δίνει κίνητρα για τη συμμετοχή ε, μειώνοντας την απόσταση που υπάρχει μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής εξουσίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε καινοτόμου τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών και για τον τρόπο χορήγηση ε, ε, πληροφοριών. Για παράδειγμα, ο Αυστριακό Συνήγορο του Πολίτη έχει κάθε εβδομάδα τηλεοπτικό πρόγραμμα με μεγάλη απήχηση. Και αυτή είναι ένα τρόπος. Αυτός είναι σημαντικό τρόπος επικοινωνία με τους πολίτες στην Αυστρία. Άλλο παράδειγμα είναι το βίντεο του Ολλανδού διαμεσολαβητή με τίτλο «Μια μέρα στη ζωή του συνηγόρου του πολίτη» που περιέχει πραγματικά περιστατικά αλλά και φανταστικά και που δίνει τη δυναμική του ρόλου του συνηγόρου του πολίτη και έτσι ενημερώνονται καλύτεροι πολίτες. Επίσης υπάρχουν κάποια φυλάδια ενημερωτικά που είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος ε, ε, για την κοινοποίηση στοιχειωδών πληροφοριών για το έργο του συνηγόρου του πολίτη και της Επιτροπής Αναφορών. Βέβαια, θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η διανομή των πληροφοριών, που είναι κάπως περιορισμένη. Θα μπορούσαν να διατίθενται και online, αλλά και έγγραφα αυτές οι πληροφορίες και καλό θα είναι να μοιράζονται σε βασικούς εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι τοπικοί φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη σύγχυση για τα πεδία δραστηριοτήτων των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε δίκτυα επικοινωνίας ε, και ε, διανομής πληροφοριών. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Διαμεσολαβητών, των Συνηγόρων του Πολίτη. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Επίσης, διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των συνηγόρων των πολιτών και των πολιτών και καλύτερη, γίνεται καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για την κοινωτική νομοθεσία. Υπάρχουν και τρόποι συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων μέσω τη Διάσκεψης των Επιτρόπων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνα και, και Κοινοβουλευτική Τεκμηρίωσης. Έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη ενημέρωση για τη διαδικασία και την επεξεργασία συγκεκριμένων αφορών. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις έχω μερικά σχόλια. Καταρχήν, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι παραβιάσει το ρωσιακού δικαίου και παραβιάσει δικαιωμάτων των πολιτών εντοπίζονται γέρος και διορθώνονται. Ίσως και μέσω των μέσων κοινωνικής ε, δικτύωσης θα μπορούσαμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό ή hashtag που να αφορά ακριβώς αυτό το θέμα. Να προωθεί δηλαδή την προσφυγή στις αναφορές ή στις καταγγελίες για να ανοιχνευτούν προβλήματα παραβίασης του ενωσιακού δικαίου. Επίσης, σε μια τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσαν να, να, να δίνονται πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές, ε, για να δίνονται κίνητρα σε άλλες χώρες να μιμηθούν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, ε, η δικτύωση μεταξύ των συνηγόρων των πολιτών και των επιτροπών αναφορών και αυτή η δικτύωση θα μπορούσε να βοηθήσει την ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Συγκέντρωση πληροφοριών, συγκέντρωση στοιχείων για τον αριθμό των αναφορών και των καταγγελιών που υποβάλλονται και τι συνέχεια δίδεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εντοπιστούν τα προβλήματα και να βρεθούν κάποιες λύσεις. Ένα αυτόνομο κεφάλαιο στις ετήσιες εκθέσεις των Επιτροπών Αναφορών ή των Συνηγορών των Πολιτών και με τέτοια ειδικά κεφάλαια σε εκθέσεις θα μπορούσαμε να προβάλλουμε όλα αυτά τα θέματα. Και επίση αυτό το κεφάλαια θα μπορούσαν να συμπληρωθούν σε μια ξεχωριστή έκθεση για αυτά τα θέματα. Και τέλο, ποιε είναι οι προτάσει για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή και μια πιο στενή επαφή των θεσμών αυτών με του Ευρωπαίου πολίτε. Καταρχήν, να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό των νέων τεχνολογιών για την διεύρυνση τη συμμετοχή. Να έχουμε συμμετοχή μέσω των κινητών τηλεφώνων, να γίνονται μέσω του βίντεο ε, οι αναφορές, ή επίσης να γίνεται αυτόματη μετάφραση των αναφορών των καταγγελιών, καλύτερη επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ε, επίσημες πλατφόρμες για να έχουμε καλύτερη επαφή με τους ε, υποβάλλοντες στην αναφορά, τους συντάκτες ε, της καταγγελίας και όλους όσους τους υποστηρίζουν. Επίσης, να γίνει καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση με κατάλληλους δείκτες, δηλαδή αφενός ε, από τη φάση της, ε, του θεσμικού σχεδιασμού, αλλά και την συμμετοχή των βασικών ε, παικτών, που είναι οι διαμεσολαβητές, οι επιτροπές αναφορές, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες. Και επίση είναι σημαντικό με συγκέντρωση πληροφοριών από τους συντάκτες των αναφορών να κάνουμε μια αξιολόγηση των εμπειριών που βίωσαν οι καταγγέλλοντες ή οι αναφερόμενοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να δίνουν δηλαδή δημοσκοπήσεις και έρευνες σε δύο φάσει: Μία έρευνα κατά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αναφορά και μία δεύτερη έρευνα στο τέλος, μετά τη διεκπαιρέωση, για να δούμε αν ανταποκρίθηκε η διαδικασία στις προσδοκίες του πολίτη ποιο ήταν, και ποιο ήταν ο αντίκτυπο που είχε η διαδικασία στην εμπιστοσύνη που έχει ο, στα θεσμικά όργανα, γιατί κάποιες μελέτες ήδη ε, δείχνουν ότι είναι θετικό ο αντίκτυπο μετά την εκπαιδεύση τη διαδικασία, αλλά δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Επίση, στοχευμένε εκστρατείε ε, σε ομάδες που είναι πιο απομακρυσμένε από τα θεσμικά όργανα. Για παράδειγμα, σύνταξη ενημερωτικών φυλαδίων. Στοχευμένων όμως προς συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Επίσης, τα φυλάδια αυτά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες και στις γλώσσες των βασικών κοινοτήτων ε, μεταναστών και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Αυτά προς το παρόν και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τυπόσια, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά σας μας ευνεύσατε και μας δώσατε μία πολύ καλή εικόνα της ε, κατάστασης. Τώρα με χαρά μου θα δώσω το λόγο στους επόμενους τέσσερις ομιλητές, τέσσερις διαμεσολαβητές από τέσσερα διαφορετικά κράτη-μέλη. Και θα ζητήσω πρώτα από την κυρία Σίλβια Σπούρεκ να λάβει το λόγο αναπληρώτρια επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Πολωνία. Και έχετε το λόγο, κυρία Σπούρεκ. Καλησπέρα σα. Θα μιλήσω αγγλικά. Σα ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και μια που μιλώ ε, από τη σκοπιά του Πολωνού συνηγόρου του πολίτη του Δ. Άνταμ Μπότναρ και από την προοπτική των, ε, του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι ανεξάρτητο ο η, η παρέμβαση μου θα είναι πιο ουσιαστική και όχι τόσο τυπική. Ε, έχουμε τα τελευταία χρόνια ότι οι νομικοί και δικαστικοί μηχανισμοί δεν είναι αρκετά αποτελεσματική και η μεταφορά του ενωσιακού δικτύου, ε, δικαίου δεν ανταποκρίνεται πολλές φορές στα δικαιώματα και στις ε, ευρωπαϊκές αξίες και δεν προστατεύονται πάντα τα δικαιώματα εθνικά όπως έχουν προβλέψει οδηγίες το ενωσιακό δίκαιο. Και για να ξεκινήσουμε, όπως ξέρουμε όλοι, οι ευρωπαϊκές οδηγίες προστατεύουν τους πολίτες των κρατών μελών κατά των διακρίσεων, αλλά μόνο περιορισμένα. Η προστασία είναι σχετικά ευρεία στην περίπτωση διακρίσεων για φιλετικούς ή εθνοτικούς λόγους. Είναι όμως ε, μικρότερη προστασία σε περίπτωση διάκρισης λόγω φύλου και πολύ περιορισμένη, πολύ περιορισμένη προστασία κατά διακρίσεων ε, ε, των ανθρώπων με αναπηρία ή των μη Όλο παραδόξου η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει άνισα του πολίτε, παρόλο ε, που οι νόμοι εξασφαλίζουν ισότιμη ε, μεταχείριση. Και μάλιστα η, ε, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει το δικαιώμα τη σχετικά. Έχουμε βέβαια ήδη τον Ιούλιο του 2008 το σχέδιο οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία όμως οδηγία δεν έχει εγκριθεί ουδέποτε. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα της έλλειψης πολιτικής βούλης των κρατών μελών, καθώς και έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τονώσει την ελληπή βούλη των κρατών μελών. Και οι επιλεκτικές πρωτοδιατάξεις της οδηγίας κατέληξαν στην υιοθέτηση ελαττωματικών εθνικών νόμων. Για παράδειγμα, ο πολωνικός νόμος για την εφαρμογή κάποιων δια... κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίση μεταχείριση. Όταν διαβάζουμε τον πολωνικό νόμο, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, για παράδειγμα, ότι οι διακρίσει κατά εθνικών, εθνοτικών μειονοτήτων σε ό,τι αφορά την πρόσβασή του στην παιδεία απαγορεύεται, αλλά η διάκριση ει βάρο άλλων πολιτών στην ίδια περιοχή λόγω γενετήσιου προσανατολισμού επιτρέπεται ή τα θύματα φυλετικών διακρίσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στο ε, σύστημα υγείας μπορεί να αντιμετωπιστεί και να αποζημιωθούν, αλλά άτομα με αναπηρίες που έχουν υποστεί επίσης άνηση μεταχείριση δεν έχουν δικαίωμα σε αποκατάσταση. Επίσης, ε, ανεπαρκή μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών στην πολωνική νομοθεσία έχει ε, εντοπιστεί στο θέμα της υλοτόμηση στο δάσος της Μπιαγοβιέσκα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολωνία έχουν υπογράψει τη σύμβαση για πρόσβαση σε πληροφορία, δημόσια συμμετοχή και στη διαδικασία λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά θέματα. Σύμβαση του όρχου. Και μάλιστα οι διατάξει τη σύμβαση του όρχου περιλαμβάνουν τι κοινοτικέ οδηγίε που απαιτούν από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε μία. Ε, ε, ε άσκηση προσφυγής σε ανεξάρτητο σώμα και αμερόληπτο προκειμένου να αφισβητηθεί μία απόφαση. Ε, στην Πολωνία όμω απαιτείται να έχουν συμμετέχει και στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αλλιώ αποκλείονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και η ασυνέπεια μεταξύ ενωσιακού και εθνικού δικαίου έχει δύο διαστάσεις στην περίπτωση του δάσου της Βιαγοβιέσκα. Καταρχήν, οι, πολυ... οι πολωνικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ δεν μπορούν να ασκήσουν έφεση η προσφυγή κατά απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνη σε ένα διοικητικό δικαστήριο. Θα μπορούσαν να κάνουν καταγγελία μόνο εφόσον είχαν, είχαν συμμετάσχει σε διαδικασίε που κατέληξαν στην έκδοση τη απόφασης. Καμία όμω περιβαλλοντική ΜΚΟ δεν συμμετείχε στις διαδικασίες αυτές. Ως εκ τούτου, ο Πολωνός συνήγορο του πολίτη προσέφηκε σε διοικητικό δικαστήριο κατά τη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο. Παρ' όλα αυτά όμω τα διοικητικά δικαστήρια και στους δύο βαθμούς έκριναν μη παραδεκτή την προσφυγή του Πολωνού συνηγόρου του πολίτη γιατί θεώρησαν ότι το αντικείμενο της καταγγελίας ήταν εκτός ε, της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων στην Πολωνία. Και αυτή είναι η δεύτερη διάσταση. Επιπλέον, τα επιχειρήματα του συνηγόρου του πολίτη στην καταγγελία του ήταν σωστά, όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ταυτόχρονα όμως, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αρνήθηκε το αίτημα του συνηγόρου του πολίτη Πολωνία Πολωνίας για τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλίσει και έλεγχο τη κοινωνία των πολιτών επί των αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, όπω ήταν η απόφαση για το δάσος Μπιαλοβιέτσκα. Τρίτον, και λυπούμε που είμαι τόσο ομοί σε αυτά που λέω, θα πρέπει να υπενθυμίσω μια κατάσταση που ήταν η λιδία αλήθω για την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των, ε, θεσμι... των νομοθετικών διατάξεων. Πρόκειται για την ε, μεταναστευτική κρίση που δημιούργησε τεράστια πρόκληση στην Ευρώπη να υποδεχθεί τεράστιο αριθμό ε, μεταναστών και προσφύγων και δυστυχώς άφησε πολλούς αβοήθητους. Η Πολωνία μετά από δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σεπτεμβρίου του 2015 δεσμεύτηκε να δεχτεί συνολικά 6.182 αλλοδαπούς υπηκόους. Και παρά τι ε, επανειλημμένε εκκλήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Πολωνία δεν τήρησε την υπόσχεσή τη και την υποχρέωσή τη. Ε, μια έλλειψη πολιτικής βούλησης κατέληξε σε σημαντική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Χιλιάδες γυναίκες, άνδρες και παιδιά έμειναν αβοήθητοι ή πνίγηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη. Ένα άλλο πρόβλημα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η άρνηση να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, σε διαδικασίες χορήγησης ε, διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς πολίτες στην Πολωνία οι ενδιαφερόμενοι από την απόφαση δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, ούτε τα πιστήρια που συνέβαλαν στη λήψη σχετικής απόφασης, ούτε έχουν ε, πρόσβαση σε ε, πραγματική έφεση ή προσφυγή με βάση τη Σύμβαση Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, πρέπει να προβλεφθεί κανονικό δικαίωμα προσφυγής, όπως ε, προτείνει το δικαστήριο, που ε, ε, αναφέρει ότι το ενδιαφερόμενο μέρος έχει, θα πρέπει να ε, ενημερώνεται για τους λόγους που στοιχειοθέτησαν την εις βάρος του απόφαση, είτε διαβάζοντας την απόφαση, είτε λαμβάνοντας ενημέρωση για την απόφαση. Αυτό είναι κάποια παραδείγματα που δείχνουν ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών δεν τη χάνουν επαρκώς προστασίας. Ο Πολωνός συνήγορος του πολίτη αντιμετώπισε όλα αυτά τα θέματα και απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές με βάση και την ομολογία του ΔΕΚ. Χωρίς όμως ισχυρή προστασία από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, ο Εθνικός Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει δυνατότητα να βελτιώσει την κατάσταση από μόνος του. Και ας μην ξεχνούμε ότι κάθε νομοθετική πράξη αφορά τους ανθρώπους, τους πολίτες, τις ανάγκες και τα όνειρά τους. Το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να λύσει τα προβλήματά τους ή και να εκδηγηθεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους ή να τους αφήσει πίσω. Είμαστε στην 16η μέρα ακτιβισμού για την αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου. Θέλουμε ειδική προστασία με βάση την σχετική οδηγία για τα θύματα, προκειμένου να καταπολεμήσουμε τη βία λογοφύλου, την ενδοοικογενειακή βία και τη σεξουαλική βία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα μπορούσα να αφιερώσω όλη μου την παρέμβαση σε αυτά τα θέματα τη βία λογοφύλου, γιατί χρήζουν εκτενού συζήτηση και εμβριθού συζήτηση και ελπίζω να έχω αντίστοιχη ευκαιρία στο μέλλον. Ω εκ τούτου, σήμερα θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η οδηγία αυτή δεν έχει μεταφερθεί πλήρως και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη επαρκώς στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βλέπετε την αντίδραση στην αίθουσα. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, με μεγάλη μου χαρά θα δώσω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, την Μαρία Πατάκιοβα είναι συνήγορος του πολίτη στη Σλοβακία. Καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες, κύριε Πατάκηβα. έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνήσαμε στο πάνελ να χρησιμοποιήσουμε τη μητρική μας γλώσσα και δεν ήταν παρούσα η συνάδελφος από την Πολωνία τότε. Τέλος πάντων, χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στη Σλοβακία. Η παρουσίασή μου θα εστιάσει στους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και είναι στην ίδια γραμμή με τα όσα ακούσαμε πριν το μεσημέρι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω λίγα λόγια για το έργο του συνήγορου του πολίτη στη Σλοβακία. Έπειτα θα περάσω στις ε, λεπτομέρειες για το μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, την σχετική ενωσυνακή νομοθεσία και την ειδική έκθεση του 2017 που παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο της ε, Σλοβακίας και τα συμπεράσματα από αυτή την ειδική έκθεση. Ο συνήγορος του πολίτη στη Σλοβακία περιγράφεται στο Σύνταγμα της ε, Δημοκρατίας της Σλοβακίας και προσθέθηκε η λειτουργία αυτή στο Σύνταγμα το 2001. Ε, βλέπετε τις αρμοδιότητες του συνήγορου του πολίτη στην Σλοβακία στη διαφάνεια αυτή. Ο θεσμός αυτός λοιπόν στη Σλοβακία είναι πάνω από 15 ετών και νομίζω πως βλέπουμε όλο και περισσότερο τα ωφέλη του συνήγορου του πολίτη στη δημοκρατία της Σλοβακίας. Τα κυριότερα στοιχεία του συνηγόρου του πολίτη είναι τα εξής. Είναι ρετός αντιπρόσωπος, εθνικός συνήγορος του πολίτη και αυτόνομο, αυτόνομος θεσμός. Επομένως, Μπορώ να πω ότι οι συνάδελφοι συνήγοροι του πολίτη στις άλλες χώρες εκπροσωπούν το, το γραφείο του συνήγορου του πολίτη, ενώ στη Σλοβακία είναι ένα πρόσωπο συνήγορο του πολίτη. Εγώ δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση, αυτή την εποχή. Περνάμε τώρα στο, στα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Στη Σλοβακία υπάρχουν 203 τέτοια εργοστάσια. θα μπορούσαν να υπάρχουν 375 παραπάνω έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν ε, το πλήρες δυναμικό των ε, ποταμών της χώρας. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε διαφορά την ύπαρξη των ε, μικρών υδροελεκτρικών σταθμών. Καταρχάς, από το πρωτόκολλο του Κιώτο απορρέει ότι οι χώρες που το επέγραψαν οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ως αποτέλεσμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία δυνατότητα είναι να χρησιμοποιηθεί η δύναμη των ποταμών για την παραγωγή ενέργειας. τα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια ε, θεωρούνται μικρά όταν ε, η παραγωγή τους δεν ξεπερνά τα τις 10 ε, μεγαβατόρες. οι επιπτώσεις των υδροηλεκτρικών εργοστασίων στο περιβάλλον είναι ε, μικρότερες από ό,τι των άλλων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Οι εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου είναι μικρότερες, το κόστος μεταφοράς είναι επίσης χαμηλότερο και επίσης ε, συνεισφέρουν στην ενεργειακή ασφάλεια και στη μείωση του κόστου σε παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, τα μειονεκτήματα είναι επίση πολλά. Αλλάζουν τη συγκέντρωση οξυγόνου στους ε, ποταμούς, αλλάζουν την ικανότητα αυτοκαθαρισμού ε, των υδάτων και επηρεάζουν την ε, χλωρίδα και πανίδα των βιοτόπων. Κατακαιρματίζουν τα αιτήματα και κινδυνεύουν μάλιστα να καταστρέψουν με πολλές περιοχές. Κατακαιρματίζεται λοιπόν η συνέχεια του φυσικού τοπίου από τα φράγματα, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την ε, μετανάστευση των ε, ψαριών και την ε, αναπαραγωγική τους ικανότητα κατά επέκταση. Τα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια θεωρούνται οικονομικά, όμως έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε αποτελεσματικά τις διάφορες μορφές ενέργειας θα πρέπει να μην παραβλέπουμε και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, στα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια υπάρχει πρόβλημα με ε, τον αποδεκατισμό του περιβάλλοντος οικοσυστήματος. Η φύση από μόνη ε, αυτορυθμίζεται. Και υπάρχει κύκλος στα οικοσυστήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα ε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας μέχρι το 2020. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου και θεωρώ ότι η οδηγία για τις μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς και η οδηγία για ε, την στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλη μια οδηγία για ε, το νερό καθώς και την ε, οδηγία για τους οικοτόπους. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος από τη μία και από την άλλη παροτρύνεται η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση ανάμεσα στις ε, οδηγίες, ανάμεσα στα νομοθετήματα και προσπάθησα εδώ να παραθέσω διάφορα άρθρα του συντάγματος της Σλοβακίας τα οποία αποτελούν τη βάση του έργου του συνηγόρου του πολίτη. Με βάση τα άρθρα αυτά διαπιστώνεται αν έχουν ε, υπάρξει παραβάσεις. Ιδιαίτερα το άρθρο 46 για το δικαίωμα πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και το σχετικό άρθρο για την νομική και ε, ενδική προστασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνήγορο του πολίτη στην ε, Σλοβακία. Σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να πούμε ότι τον Μάρτιο του 2017 η ηθική έκθεση ανέφερε αυτά τα συγκρόμενα συμφέροντα. Το να παράγεται δηλαδή από τη μία ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ και από την άλλη να ε, γίνονται σεβαστά τα πρότυπα προστασία του περιβάλλοντο. Η έκθεση λοιπόν υπευλήθη στο Κοινοβούλιο και στο Εθνικό Συμβούλιο της ε, Σλοβακίας το 2017 οδήγησε σε μία, στη σύσταση μιας ε, εξεταστικής επιτροπής από το συνήγορο του πολίτη, διότι υπήρχαν πολλές καταγγελίες από τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές εφάρμοσαν τις ε, προαναφερθήσεις οδηγίες. Στόχος ήταν να γίνει αξιολόγηση για το αν οι αποφάσεις συμμορφώνονταν με την εθνική νομοθεσία και αν αυτή η συμμόρφωση ήταν επίσης συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο. Το πόρισμα της Επιτροπής αυτής ήταν ότι έχουν σημειωθεί σοβαρές παραβιάσεις ε, της νομοθεσίας αλλά και των ε, βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι πολίτες δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς ούτε και μπορούσαν να ασκήσουν ε, τα δικαιώματά τους σε ό,τι φορά τα ένδικα μέσα. Οι παραβιάσεις ήταν συστηματικές. Βλέπαμε να επιμένουν τα ίδια προβλήματα. Πέραν αυτών, οι αρχές, χρησιμοποιώντας φορμαλιστικές μεθόδους, και χωρίς καθόλου συνέπεια στην ε, επιλογή τους, δρούσαν αυθαίρετα. Είχαν στόχο τη, την παραγωγή ενέργειας ε, παραβλέποντας και αγνοώντας εσκεμένα του, την περιβαλλοντική καταστροφή. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αποτυχία συνεκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν παταγώδης, καθώς και η εφαρμογή των ε, οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Μία από τις ε, υποθέσεις που αναφέρει η έκθεση είναι ένα εργοστάσιο στο ΝΤΕΚΟ. Εκεί υπάρχει μία ειδοποίηση για ε, παραβίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το, 2, το Νοέμβριο του 2014. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα εργοστάσια στον ίδιο ποταμό, τα οποία αθρηστικά οδηγούν στην επιδείνωση της ποιότητας του νερού και του βιοτόπου, η καταστροφή συνεχίζεται. Υπάρχει, ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας το οποίο χρησιμοποιεί νερό και στη συνέχεια το απελευθερώνει στον ε, ποταμό. Άλλο παράδειγμα, το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη Σάλκοβα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση του χωριού, σε απόσταση 20 μέτρων από σπίτια έχει οδηγήσει σε διάφορες ε, ζημιές. Οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν από την ηχορύπανση ε, και από ηχορύπανση χαμηλών συχνοτήτων που προκαλεί το εργοστάσιο αυτό. Το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη είχε ως εξής. Χρειάζεται στρατηγικός ε, σχεδιασμός έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα συνολικός κατάλογος των ε, επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ύπαρξη αυτή των ε, μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων, ο οποίος με τη σειρά του θα χρησιμοποιηθεί κατά τη, διάρκεια, κατά διαδικασία αδειοδότησης για την κατασκευή αυτών των εργοστασίων. Επίσης, χρειάζεται αύξηση της διαφάνειας στην όλη διαδικασία εντοπισμού των ε, ποταμών εκείνων όπου υπάρχει δυναμικό παραγωγής υδροελεκτρικής ενέργειας. Όταν έγινε η σύνταξη της έκθεσης δεν είχαμε διαθέσιμα δεδομένα τέτοιου τύπου. Και οι πληροφορίες αυτές ήταν στα χέρια μίας ε, εταιρείας η οποία βρισκόταν ε, υπό κρατική διαχείριση. Θεωρώ ότι τα σχέδια για την ε, δυνατότητα χρησιμοποίησης υδροελεκτρικής ενέργειας ε, της ε, Σλοβακίας δεν περιείχαν τις συστάσεις από την αξιολόγηση των αθρηστικών επιπτώσεων των υδροελεκτρικών εργοστασίων. Επίσης, τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επικαιροποιηθεί, δεν έχουν τροποποιηθεί για να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις και η πρόταση του 2013 δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θρηστικά, αυτές οι θρηστικές επιπτώσεις. Έγινε προσφυγή λοιπόν στο δικαστήριο για το ε, αναθεωρημένο αυτό έγγραφο. Η δίκη συνεχίζεται ακόμα. Συμπερασματικά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ζωτική σημασίας να αξιολογηθούν τα ωφέλη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε, απέναντι στο, στην περιβαλλοντι... στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μόνο τότε θα πρέπει να ε, λέμε ότι ένα εργοστάσιο παράγει πραγματικά πράσινη ενέργεια πολλοί απλοί πολίτες, οι ενώσεις, οι διαφορές οντότητες που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης ε, άδεια ζήτησαν ε, ε, περισσότερη διαφάνεια. Οι ενώσεις όμως των πολιτών δεν είχαν την δυνατότητα αυτή, δεν απέκτησαν ποτέ πρόσβαση στην διαδικασία. Και στο μέλλον η νομοθεσία είτε στη Σλοβακία είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τα εξή χαρακτηριστικά. Θα πρέπει καταρχάς να ποσοτικοποιεί τα συμφέροντα και από τις δύο πλευρές, να, να ζυγίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, να αξιολογεί την ποιότητα των ε, διαθέσιμων πληροφοριών, και να μην λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη. Διότι δεν γίνεται να αξιολογήσεις ε, αυτά τα στοιχεία χωρίς τα κατάλληλα έγκυρα ε, δεδομένα και χωρίς να ακολουθηθούν αυτές οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Σάξολιν από την Φιλανδία. Είναι διαμεσολαβήτρια στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη των κοινοβουλίων, ο ρόλος του διαμεσολαβητή στη Φιλανδία είναι να παρακολουθεί την δημόσια διοίκηση προκειμένου να έχει τη βεβαιότητα ότι όλοι συμμορφώνονται με τον νόμο και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Κάνοντας κάτι τέτοιο, αυξάνουμε την εμπιστοσύνη στην δημόσια διοίκηση και στη δημοκρατία και στηρίζουμε το κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας προκειμένου να πάρω το λόγο. Αυτό που θα ήθελα να κάνω στην ε, σημερινή συνεδρίαση είναι να σας εξηγήσω τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ενωσιακό δίκαιο υπήρξε πρόβλημα στη Φιλανδία. Υπήρξα μια σειρά από αναφορές για θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και τα θέματα αυτά λήφθησαν υπόψη και από την ε, Διαμεσολαβήτρια και από τα κοινοβούλια. Πιστεύουμε ότι το θέμα αφορά πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά επειδή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα δεν είναι πάντοτε νομικού χαρακτήρα, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Ενδεχομένω έχουμε να κάνουμε με τα ίδια πράγματα, αλλά από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το πρώτο μου παράδειγμα αφορά την πρόσβαση στους, ε, στα εστιατόρια των ε, ε, τρένων για άτομα με κινητικά προβλήματα. Διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν προαπαιτούμενο στα βαγκόν ρεστοράν να έχουν ε, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα με ειδικέ ανάγκες, σε αναπηρικά μαξίδια δηλαδή. Αυτό ήταν ένα θέμα κοινοτικού δικαίου και περιορισμού του ανταγωνισμού. Συνεπώ ο διαμεσολαμητή ε, δεν μπόρεσε να λάβει μια τελική απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, όλους όσους έχουν σχέση με το, τους σιδηροδρόμους, έτσι ώστε όλοι να τη κάνουν τις ίδιες μεταχείρισεις. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορά ε, σχετικά με μια χώρα μέλος. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση Το θέμα είναι τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα από ένα άλλο κράτος μέλος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρξε, υπήρχε παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου, παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, το ότι απαιτεί το η καταβολή όλων των φόρων της περιπτώσεις που το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Οι συγκεκριμένες χώρες ήταν η Φιλανδία και το, ε, η Ολλανδία. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ήταν παράνομο αυτό που έκανε η Φιλανδία και ζητήθηκε από τον ε, Υπουργό να ευθυγραμμίσει το φιλανδικό δίκαιο με αυτό της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο παράδειγμα μου αναφέρεται στην εφαρμογή της γενικότερης αρχής του κράτους δικαίου. γενικές αρχές εφαρμογής του κράτους δικαίου από την διοίκηση. Αφορά ιδιαίτερα την αναγνώριση των ε, τυπικών προσόντων, επαγγελματικών ε, προσόντων. Η Ομποσπαν διαπίστωσε ότι οι φιλανδικές αρχές είχαν δράσει σωστά διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχε προαπαιτούμενο, δεν ήταν απαραίτητο να τύχει αναγνώρισης ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσώνο. Αλλά οι αρχές δεν είχαν λάβει υπόψη τους τις γενικέ ενωσιακέ αρχές. Εδώ και πάλι έχουμε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναφέρεται στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι νομικές αρχές, ευρύτερες νομικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εφαρμόζεται το ε, ενωσιακό δίκαιο. Το επόμενο παράδειγμά μου αφορά την εθνική νομοθεσία. Ο Κακιαδιέλων ανέφερε ότι η νομοθεσία ήταν σε φάση προπαρασκευής στη Φιλανδία και αυτό αφορούσε το θέμα του κυνηγιού. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η νομοθεσία δεν συμμορφώθηκε με τα απαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, ο διαμεσολαβητής διαπίστωσε ότι δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί δικαστική απόφαση σε, περίπτωση, σε μια περίπτωση που αφορούσε την πυκνότητα του ζωικού βασιλείου και ότι σε τελική ανάλυση είναι θέμα των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ένα περαιτέρω παράδειγμα που αφορά τις ε, συνταγματικές αρχές ε, της ε, χρηστής διαχείρισης καθώς και το θέμα της διαφάνειας και της έγκαιρης διοικητικής δράσης. Το θέμα αυτό αφορά την εφαρμογή του νοσιακού δικαίου στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Η καταγγελία ήταν ότι ο καταγγέλων δεν είχε λάβει πληροφορίες από τις αρχές ασφάλειας τροφίμων, ασφάλειας τροφίμων. Οι αρχές ασφάλειας τροφίμων απήντησαν ότι υπήρχε έλλειψη σαφήνεια σχετικά με την ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου και η Εθνική Αρχή της Φιλανδίας αναζήτησε την άποψη άλλων κρατών μελών καθώς και της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό αφορούσε το δικαίωμα στην ενημέρωση. σε σχέση με το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα. Ο καταγγέλων, ε, μάλλον ο διαμεσολευτής αναγνώρισε ότι η αρχή αναζήτησε πληροφορίες από αλλού, αλλά χρειάστηκε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αρχή θα έπρεπε να έχει υιοθετήσει μία απόφαση σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε το θέμα να ε, είχε εκδικαστεί ενώπιον δικαστηρίου και θα χρειαζόταν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί. Το τελευταίο μου παράδειγμα αφορά το απαιτούμενο, το προαπαιτούμενο εμπορικής ε, πίστης. Στη συγκεκριμένη παράπτωση, περίπτωση η καταγγελία αφορούσε το χρόνο που απαιτήθηκε από το τελωνίο για να ε, εκτελωνήσουν εισαγόμενα αγαθά. Είπαμε, ε, ο, ο είπε ότι η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να ενεργεί ταχαίως και να εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών δίχως αντικειολόγητη καθαστήριση. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Έχω δύο σημεία που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα. Το πρώτο φορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων διαπίστωσα ότι με τη μετακίνηση στην ε, αποφάσει με βάση την πλειοψηφία, η εφαρμογή του κοινωτικού του νοσιακού δικαίου έγινε πιο δύσκολη. Ιδιαίτερα έγινε δύσκολο Κατέστη δύσκολη η επίτευξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον ίδιο το θεσμό του διαμεσολαβητή. Όταν εφαρμόστηκε στη Φιλανδία η, ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, παρατηρήσαμε ότι ο αναγκαίος μηχανισμός παρακολούθησης ή ελέγχου απαιτούσε από τον διαμεσολαβητή να γίνει επίση αντικείμενο παρακολούθησης. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Φιλανδίας, ο διαμεσολαβητής είναι υπεύθυνο για την εποπτεία όλων των δημοσίων φορέων, ακόμα και σε θέματα προστασίας του κοινού. Στο μέλλον, συνεπώς, όταν συντάσσεται νομοθεσία για θέματα όπως η προστασία δεδομένων, δεν θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την άποψη του δικαστηρίου. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και την ιδιάζουσα θέση του διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο επόμενος ομιλητής, η επόμενη ομιλήτρια είναι από την Πορτογαλία, κύριε ή κυρία Τερέζα Τανίνιο. Ανζίνιο. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους για τη συμμετοχή σας και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ε, λόγω του προχωρημένου της ώρας δεν θα επεκταθώ, θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση στη δημόσια αυτή ακρόση και του Πορτογάλου συνηγόρου του πολίτη. Όπως ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στο δίκαιο για να εξασφαλίσει την συγκεκριμενοποίηση των πολιτικών και προτεραιοτήτων της στα κράτη-μέλη. Ε, στόχος της είναι η δημιουργία μιας ισχυρότερη Ένωση. και γι' αυτό είναι αναφίβολο ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε την ομοιόμορφη εφαρμόγη του ενωσιακού δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Και Φυσικά, αναπόφευκτα εξαρτώμαστε από μια ποιοτική νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ε, την αποτελεσματικότητα σε επίπεδο εφαρμογής, εκτέλεσης ε, και τήρησης. Ε, είναι αναφυσβήτητο ότι λόγω της φύση, ο θεσμός του σφίστου, ο θεσμός του συνηγόρου του πολίτη είναι πολύ σημαντικός, έχει στρατηγική σημασία σε αυτή την κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Στην Πορτογαλία ο συνήγορος του πολίτη από το 1999 είναι ε, μαζί με τον Εθνικό Θεσμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πλήρη συμβατό με τι αρχέ των Παρισίων και ω ε, πρωταρχική λειτουργία έχει την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων ελευθεριών εγγυάται τα ε, ένομα συμφέροντα και θεμητά συμφέροντα των πολιτών και εξασφαλίζει ε, την ε, δικαιοσύνη και την νομιμότητα στην άσκηση των δημοσίων εξουσιών. Οπότε η αξία της δικαιοσύνης προηγείται της αξίας της νομιμότητας. Και όπως είπαμε και πριν από λίγο, αυτό είναι και η βασική πρόκληση των συνηγόρων του πολίτη. Να εξασφαλίσουν δηλαδή την ισορροπία ε, γιατί μπορούν να ξεπεράσουν το νόμο και μπορούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ της νομιμότητας και της σκοπιμότητας της συγκεκριμένης δράσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακριβώς αυτό το πλαίσιο, δηλαδή ο συνήγορος του πολίτη, ο συγκοιητής ε, και θεματοφύλακας ε, των δικαιωμάτων των πολιτών και στην πρόθεση και την προστασία και σε ό,τι αφορά ή παραλήψης των δημοσίων φορέων, ε, θα πρέπει να ασκεί αυτό το ρόλο του εγγυητή των, δοκιμά... των δικαιωμάτων των πολιτών και, και φυσικά ε, είναι και εγγυητής του ενωσιακού δικαίου. Γιατί με τη διπλή αυτή ιδιότητα και με πολλούς παραλληλισμούς, ο συνήγορος του πολίτη ε, και χάρη σε μια αποτελεσματική συνεργασία και χωρίς καμία αλληλεπίδραση λειτουργική ή θεσμική, ασκεί τα καθήκοντά του και συνεργάζεται φυσικά και με τον Ευρωπαίο Διαμοσιολαβητή. Ε, και ε, νομίζω ότι δεν είναι περιττό να τονίσουμε ότι σε αυτή τη διάσκεψη η το θέμα που είναι η εφαρμογή του δικαιώματος ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό να ε, συναρτήσουμε τη λειτουργία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε συνδυασμό με τους ε, εθνικούς συνηγόρους του πολίτη. Έτσι θα πραγματοποιήσουμε αυτή την συμμετοχική έννοια της ηθαγένειας και θα βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να εφαρμόσουν καλύτερα το ενωσιακό δίκαιο. Και φυσικά να προστατεύσουμε τους πολίτες όταν προσκρούσε εμπόδια σε ό,τι αφορά την ε, σωστή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήθελα να σας ενημερώσω για το ρόλο του συνηγόρου του πολίτη στην Πορτογαλία και πώς ασκεί τη λειτουργία και τα καθήκοντά του. Φυσικά ενημερώνει τον πολίτη για τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και αυτός είναι θεσμικός ρόλος ε, και γι' αυτό έχει πολλά μέσα στη διάθεσή του. Ε, στη διάρκεια της ζωής του, ε, ο συνήγορος του πολίτη υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβάνοντας αυτά αρχές, κανόνες και διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο. Και ακριβώς με τη συγκεκριμένη αυτής της ε, προσέγγισης οργανώσαμε διασκέψεις, εκστρατείες, ενημερωτικές δράσεις και των δημοσίων αρχών, των, ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ε, υπηρεσιών ασφαλείας, των δικαστικών, ακόμη και των της παιδείας. Προσπαθούμε να φτάσουμε στους πάντες και μάλιστα χρησιμοποιώντας εύληπτη διατύπωση, μια ορολογία κατανοητή, γιατί είναι σημαντικό οι θεσμικοί φορείς που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες ε, να επικοινωνούν εύκολα με τους πολίτες και μάλιστα με αποκεντρωμένο τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει να αποφύγουμε τη συγκέντρωση του έργου, του έργου μας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα πρέπει να μπορούμε να φτάσουμε και στην Εδωχώρα και στην Ήπεθρο και ακόμη και στην ψηφιακή αυτή εποχή λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό ψηφιακό αλφαβητισμό που παρατηρείται σε ορισμένες χώρες. Πρόθεση των δικαιωμάτων σημαίνει και πρόληψη, σημαίνει καλύτερη συνειδητοποίηση, σημαίνει προσπάθεια μείωσης του κενού και του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των δημόσιων πολιτικών και των πολιτών, που υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να φέρουμε το νόμο που διέπεται από κάποιες αξίες ε, σε επαφή με την κοινωνία, που μερικές φορές έχει διαμετρικά αντίθετες αξίες. Και αν θέλουμε ποιοτική ε, νομοθεσία, δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στην απλή θέσπισή τη ή στην απλή μεταφορά των οδηγιών. Σημαντικό στοιχείο είναι στην εφαρμογή η εξασφάλιση και η διάδοση και της γνώσης, εξασφαλίζοντας ε, ότι το δικαίωμα θα απομακρύνεται από ένα θεωρητικό πρόγραμμα και θα ε, μετουσιώνεται σε ένα πρόγραμμα δράσης. Είναι αλήθεια βέβαια ότι στη δράση του συνηγόρου του πολίτη της Πορτογαλίας ε, μεγάλη έμφαση δίνουμε στην ε, λήψη και επεξεργασία των καταγγελιών. Δεν έχουμε στοιχεία για τον αριθμό των καταγγελιών στους οποίους ο καταγγέλων επικαλείται το ενωσιακό δίκαιο. Πάντως, όταν ε, μια καταγγελία αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, οι καταγγέλλοντες ε, επικαλούνται το πορτογαλικό σύνταγμα που πέραν των συνταγματικών αρχών περιλαμβάνει και έναν εκτενή κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βέβαια, από τη στιγμή που ο συνήγορος του πολίτη δεν δεσμεύεται από τα επιχειρήματα που ε, παρουσιάζουν οι καταγγέλλοντες στις αιτιάσεις τους, μπορεί να επικαλεστεί το ενωσιακό δικαίωμα όταν το κρίνει εφαρμοστέο ή σχετικό με την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Και αυτό συνέβη ε, επί σειρά ετών ε, ανάλογα με την περίπτωση. Ε, έτσι συμβάλλουμε και σε μια παιδαγωγική προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την ομοιόμορφη εφαρμογή και την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Σε ό,τι αφορά τη διάκριση λόγω ηλικία, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα, ασχοληθήκαμε στην Πορτογαλία με τα ανώτατα ηλικιακά όρια εισαγωγή σε κάποιες επαγγελματικές σταδιοδρομίες ή τις διαφοροποίησεις που υπάρχουν στο πέρασμα ε, στη διαθεσιμότητα λόγω ορίων ηλικία των διπλωματικών υπαλλήλων. Το, δικαίωμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η σχετική νομολογία του ΔΕΚ στις περιπτώσεις αυτές έχουν τεράστιο βάρος και συνέβαλαν και η νομολογία και το νοσιακό δίκαιο στη διαμόρφωση θέσεων που θα μπορούσα να τη συνοψίσω σε εξής. Δέχονται ε, απριόρι ότι ο στόχος ε, των ε, νομοθετικών διατάξεων είναι νομότυπος και γι' αυτό σε συγκεκριμένα επαγγέλματα καλούμε την κυβέρνηση να ξανασκεφτεί τις νομοθετικές λύσεις και να βρει προτάσεις που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης. βέβαια, δεν ξεπερνάμε τα όρια μας ε, σε ό,τι αφορά τα ηλικιακά όρια. Θα πρέπει πρώτα να διαπόμεστε από τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και φυσικά να ελέγχουμε μονίμως και να παρακολουθούμε την τήρηση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, είχαμε επίσης μια πρόσφατη νομοθετική αναθεώρηση που ε, εκπορέθηκε και πάλι από το Ενωσιακό Δίκαιο και αφορούσε μια περίπτωση αντίστροφης διάκρισης Όπω συμβαίνει όταν μια χώρα αντιμετωπίζει δυσμενώ του υπηκόου του σε σχέση με τη μεταχείριση των υπηκών άλλων χωρών μελών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια διόρθωση που έγινε χάρη σε μια νομοθετική αναθεώρηση, η περίπτωση αφορούσε τους πολιτικούς μηχανικού, μηχανικούς που λόγω της κατάρτισης που είχα στην ε, Πορτογαλία δεν μπορούσαν να συνεχίσουν κάποιες δραστηριότητες και στον τομέα της αρχιτεκτονικής, κάτι που στο παρελθόν επιτρεπόταν και σε άλλες χώρες θα εξακολουθούσε να επιτρέπεται χάρη σε μια οδηγία που μετέφεραν άλλες χώρες μέλη στην ιστορική του ένωμη τάξη. Επίσης, σε τέτοια περίπτωση θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, μια άλλη καταγγελία που οδήγησε σε, σε νομοθετική αναθεώρηση. Αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στις δημόσιες παιδικές χαρές και αφορούσε θέματα ε, ενιαίας αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο συνήγορος του πολίτη ε, επέσει την προσοχή του νομοθέτη όχι μόνο στην ε, ε, εθνική εφαρμογή αυστηρότερων διατάξεων που δεν αύξαναν ταυτόχρονα την ασφάλεια των παιδιών, αλλά στην ανάγκη ε, λόγω των τεχνικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας να κοινοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ε, νομοθετικές τροποποιήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των κανόνων. Τώρα, σε ένα άλλο πλαίσιο και για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να σας μιλήσω για μια άλλη κατηγορία καταγγελιών, όπου ο συνήγορος του πολίτη μπορεί στην Πορτογαλία να διαδραματίσει έναν παιδαγωγικό ρόλο. Ε, δικαιολογεί και εξηγεί τη σημασία που έχουν κάποιες νομοθετικές διατάξεις που απορρέουν από τη μεταφορά ε, κοινοτικών οδηγιών όταν οι πολίτες δεν το αντιλαμβάνονται έτσι. Αυτό συνέβη, συμβαίνει συχνά όπως θα φαντάζεστε με την περιβαλλοντική νομοθεσία και κυρίως ε, με την ατμοσφαιρική ε, ρήπαση. Για παράδειγμα, πολύ συχνά οι πολίτες αμφισβητούν κάποια περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία των οχημάτων ε, στα κέντρα των πόλων. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μας να αποκαταστήσουμε την αντίληψη της ισορροπίας των αξιών που διακυβεύονται εδώ και να διαπαιδαγωγήσουμε τους πολίτες για το πόσο σημαντική αξία είναι το περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος και να ενημερώσουμε τον πολίτη για τη σχέση που έχει το περιβάλλον με την αρχή της αηφόρου ανάπτυξης, κάτι που δεν τι βλέπει συχνά ο Ευρωπαίος πολίτης, αυτή τη συσχέτιση. Επίσης, ε, φυσικά πολλά εξαρτώνται από την ε, εφαρμογή των ε, ενωσιακών κανόνων. Γι' αυτό θα πρέπει να αναγόμαστε συνεχώς στο ενωσιακό δίκαιο και στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό κάνουμε στην Πορτογαλία και στην ε, Πορτογαλία δεν είμαστε απλοί με διαμεσολαβητές, αλλά ταυτόχρονα και Εθνικό Ινστιτούτο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και βασικός φορέας για την εφαρμογή της σύμβασης ε, για τη... κατά των βασανιστήριων. Και έτσι ενημερώνουμε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συστήματος και σίγουρα η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είναι χαρακτηριστικό δείκτη αποκεντρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή στι εσωτερικέ έναμε τάξει. Ε, και μπορώ να ε, τονίσω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προ ένα πιο συνεκτικό σύστημα προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότητα απέναντι στα δικαιώματα ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, πιστεύω αναφίβολα ότι ο δρόμος μπροστά μας θα είναι μακρύς και θα πρέπει να ενδύνουμε τις δράσεις μας και σε επίπεδο πρόθεσης και σε επίπεδο προστασίας. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων ε, για καλύτερη ανταλλαγή εμπειριών και των πρακτικών. Και πολύ σημαντικό επίσης θέμα είναι η παρακολούθηση, γιατί έχουμε επίγνωση της σημασίας που έχουν ε, οι πληροφορίες και τα στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε το θεμελιώδες βήμα προς πιο ποιοτικέ δημόσιε πολιτικέ. Ευχαριστώ. Thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν και το τέλος των ε, παρουσιάσεων. Τώρα θα δώσω το λόγο σε εσάς και ήδη έχω λάβει έτοιμα ε, από τον κύριο Ρόμπερτ Μάματο από την ε, Πολωνική Γερουσία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έφυγε η Πολωνέζα συνήγορος του πολίτη για να σχολιάσω τα λεγόμενά της. Ε, στην Πολωνική Γεωρουσία έχουμε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου και στην Επιτροπή αυτή κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να υποβάλει καταγγελίες, να ασκήσει προσφυγή, να υποβάλει αναφορά για να διορθωθούν διατάξεις ε, ή να καταγγείλει κάποιες παραβιάσεις. Και ακόμη και ιδιώτης μπορεί να απευθυνθεί σε αυτή την Επιτροπή της Πολωνικής Γερουσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ομάδες πολιτών. Τώρα, τι θέματα πραγματεύεται η Επιτροπή Αναφορών και Δικαιωμάτων του Πολίτη. Ελευθερία έκφραση και συνείδηση, προστασία τη υγεία, τα δικαιώματα των ανηλίκων, ε, η σύνδεση του, βουλευτικού, με το... Ε, της βουλευτικής έδρας με την έδρα του γερουσιαστή, ε, θα, δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε, εργατικό δίκαιο, θέματα ραδιοτηλεόρασης, δικαιώματα του καταναλωτή, δικαιώματα ιδιοκτησίας. Το, η Επιτροπή Αναφορών Κράτους Δικαίου και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων λαμβάνει πολλές αναφορές από τους Πολωνούς πολίτες και πολύ συχνά εμ, κάνουμε εισήγηση για νομοθετική αναθεώρηση. Η συνήγορος ε, του πολίτη στην Πολωνία έχει πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Αναφορών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βέβαια, η Επιτροπή της Πολωνικής Γερουσίας έχει τα δικά της καθήκοντα και ο συνήγορος του πολίτη στην Πολωνία έχει τα δικά του καθήκοντα. Πάντως, σίγουρα με αγαστή συνεργασία υλοποιούμε καλύτερα τους στόχους μας. Και στον ε, Πολωνό Διαμεσολαβητή, στον Πολωνό Συνήγορο του Πολίτη, απευθύνεται ε, άμεσα ο ιδιότητας για θέματα πολύ πιο ατομικά. Ενώ η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Πολωνικής Γερουσίας ε, ασχολείται με πιο γενικά θέματα γιατί μπορεί να εισηγηθεί και νομοθετική αναθεώρηση. Ενώ ο διαμεσολαβητής μόνο συστάσεις μπορεί να κάνει. Βέβαια, δεν είναι πάντα η συνεργασία με τον Πολωνό διαμεσολαβητή ιδεώδης και πάντα υπάρχει δυνατότητα για βελτιώσεις και σε αυτό προσβλέπουμε. Πάντως, ως Επιτροπή Αναφορών από ε, κράτους δικαίου και ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο του διαμεσολαβητή. Ο συνήγορος του πολίτη στην Πολωνία πραγματικά κάνει πολλά για τη βελτίωση της εφαρμογής των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην Πολωνία. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο για την υπερμετρή υλοτομία στο δάσος Μπιαλοβιέτσκα. Όπως είπε και η συνήγορος του πολίτη από την Πορτογαλία, ε, στόχος μας είναι η υποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης. Παρόμοιο πρόβλημα ε, με την ε, διαχείριση των δασών έχει και η Γερμανία. Και εκεί γίνεται προληπτική υλοτομία όπως στην Πολωνία. Για τη Γερμανία όμως κανένας δεν λέει κουβέντα. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η ισότιμη μεταχείριση την οποία όλοι προσβλέπουμε. Και φυσικά σταματήσαμε τελικά αυτή την προληπτική υλοτομία. Δεν κάνουμε τέτοια προληπτική πια υλοτόμηση στο δάσος Μπιαλοβιέτσκα, γιατί επενεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεχτήκαμε τι συστάσεις τη. Αλλά μακάρι να υπήρχε ισότιμη μεταχείριση και των χωρών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ και την Επιτροπή μας και βεβαίως τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και όσους συμμετείχαν σε αυτή την ε, ημερίδα. Ένα μεγάλο μέρος της το παρακολούθησα από το γραφείο μου, δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω εδώ. Αλλά αυτό που ήθελα να θίξω από την πλευρά μας είναι, μιλούμε για τα δικαιώματα των πολιτών και θα ήθελα να μιλήσω για τα δικαιώματα των βουλευτών διότι και οι βουλευτές είναι πολίτες, αλλά βεβαίως οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με την προβολή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι κάτι το οποίο έχω πει αρκετές φορές στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή Αναφορών. Απλά θα το πω και σε αυτή τη συνάντηση, μια και υπάρχουν ε, βουλευτές από, όλα, από αρκετά κράτη-μέλη και αντιπροσωπείες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την δικιά μας περίπτωση, με την Ελλάδα, αντικειμενική ενημέρωση. Δεν υπάρχει πλουραλισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν υπάρχει και προβολή του έργου των Ευρωβουλευτών ισότιμα. Εγώ ανήκω στο ECR που είναι η τρίτη σε δύναμη πολιτική ομάδα και εάν δείτε το καθημερινό δελτίο το οποίο εκδίδει το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα που δείχνει και μάλιστα στα αγγλικά ποια η συμμετοχή των ευρωβουλευτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα δείτε ότι η δικιά μας περίπτωση του ECR και η δικιά μου προσωπικά είναι εξασθενημένη. Θα έλεγα επί της ουσίας έχει εξαφανιστεί. Δεν μας δίνουν το δικαίωμα να προβληθούμε ισότιμα ή ως τρίτη πολιτική δύναμη στην κρατική τηλεόραση. Η κρατική τηλεόραση έρχεται εδώ στις Βρυξέλλες, έρχεται στο Στρασβούργο, χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το στούντιο και όμως η δική μας συμμετοχή και αναλογία είναι ελάχιστη. Άλλο θέμα αφορά την ιδιωτική τηλεόραση, όπου τα μεγάλα συστημικά κανάλια μας έχουν κυριολεκτικά εξαφανίσει. Επομένως μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα. Υπό ποιου όρου θα πάμε στις ευρωεκλογέ και πώς θα υπάρχει η αντικειμενική ενημέρωση, η πληροφόρηση, ο πλουραλισμός όταν επί τέσσερα και πλέον έτη μας έχουν εξαφανίσει και όταν τον τελευταίο μήνα προφανώ θα μα δώσουν ισότιμο χρόνο. Αλλά τι να το κάνει κανεί τον τελευταίο μήνα όταν επί 4,5 σχεδόν 5 χρόνια δεν έχουμε τη δυνατότητα προβολή. Και επιπλέον γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι ότι είμαι ο πρώτο σε ομιλίε και παρεμβάσει στου 751 ευρωβουλευτέ. Ακόμη και αν έκριναν με αυτό το κριτήριο θα έπρεπε η δικιά μα προβολή να υπάρχει. Θα σας αποστείλω κύριε Πρόεδρε ενδεικτικά τα δελτία τα χτεσινά και των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα για να δείτε την έλλειψη προβολής γιατί εκεί αναφέρεται σε ποια κανάλια και ραδιόφωνα βγήκαν οι ευρωβουλευτές και θα δείτε ότι μας έχουν εξαφανίσει. Εγώ ρωτάω, μπορούμε να πάμε ισότιμα στις ευρωεκλογέ. Αυτό είναι ερώτηση καθοριστική, αφορά ενδεχόμενα και άλλες χώρες, αλλά εγώ αυτό το θέτω για την Ελλάδα και πλέον δεν ξέρω σε ποιο όργανο να αποτανθώ. Να αποτανθώ στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, να αποτανθώ στην Επιτροπή Αναφορών. Το έχω θέσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έχω πει στην Κομισιόν. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει μέτρα τουλάχιστον από τώρα και για πέντε μήνες να υπάρχει προβολή των απόψεών μας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χωσέμπα Κερετσέα από την Ισπανία. Έχετε το λόγο. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Στην Ισπανία η κατάσταση είναι παρόμοια με αυτή που μας περιέγραψε η συνήγορος του πολίτη από την Πορτογαλία. Γιατί ο συνήγορος του πολίτη οργανικά υπόκειται στη Βουλή. Γι' αυτό έχουμε μεικτή αντιπροσωπεία από τη Βουλή και τη Γερουσία. Γιατί σε κοινή ε, επιτροπή, μεικτή επιτροπή Βουλής και Γερουσίας ε, είναι υπόλογος συνήγορος και όπως είπε και η πρόσωπος της Πορτογαλίας, ο συνήγορος του πολίτη είναι ο θεσμός που εγγυάται και την εφαρμογή του μηχανισμού κατά των βασανιστήριων. Υπάρχει και αυτή η αρμοδιότητα στο ρόλο του συνηγόρου του πολίτη. Επίσης, ο συνήγορος του πολίτη κάθε έξι μήνες ή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα πρέπει να λογοδοτεί επίσημα μπροστά στην Ισπανική Βουλή, στα δύο σώματα της Ισπανικής Βουλής. Και οι βουλευτές και οι γερουσιαστές που συμμετέχουν σε αυτή τη μεικτή επιτροπή των δύο σωμάτων, εκτός του ότι ζητούν από το συνήγορο του πολίτη να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις πολύ σημαντικές και να παρακολουθήσει κάποια σημαντικά ζητήματα. Πολλές τέτοιες ενέργειες ξεκινούν από πρωτοβουλία του συνηγόρου του πολίτη. Εμείς μιλούμε από τη σκοπιά του, της νομοθετικής εξουσίας που ελέγχει εντό εισαγωγικών το θεσμό του συνηγόρου του πολίτη. Αναφέρθηκαν και πολλά παραδείγματα. Στην Ισπανία ο συνήγορος του πολίτη είχε τεράστια προσφορά σε ό,τι αφορά την παρατήρηση και την εποπτεία ε, των κέντρων υποδοχής ε, παράνομων παράτυπων μεταναστών ή των κέντρων ε, παροχής ασύλου στους ασυνόδευτους ενηλίκους. Η Μεσόγειος και η Ισπανική επικράτεια είναι σημαντικές πύλες εισόδου μεταναστών και προσφύγων και ε, η παρατήρηση της ε, λειτουργίας των δημοσίων αρχών τα κέντρα αυτά υποδοχή μεταναστών ε, εξασφαλίζεται από το συνήγορο του πολίτη. Φυσικά σε κάθε χώρα ίσω υπάρχουν μικρέ διαφορέ, Πάντως ο έλεγχο και η δυνατότητα που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια απέναντι σε θεσμού όπω το διαμεσολαβητή του συνήγορου του πολίτη είναι απαραίτητα για να δούμε πόσο μέσω αυτού του θεσμού φτάνουν ε, στις δημόσιες αρχές τα παράπονα των πολιτών, οι αιτιάσεις τους, οι καταγγελίες τους, οι αναφορές τους. Ευχαριστώ πάντως για τη διοργάνωση αυτή και ευχαριστώ και όλους τους εκπροσώπους ε, των θεσμών του συνηγόρου του πολίτη που μίλησαν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γερόσοφ Βαγουένς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με ενέπνευσε ο κύριος Μαριά ε, και γι' αυτό ζήτησα και εγώ το λόγο όταν ε, μίλησε για πλουραλισμό και για έλλειψη πρόσβασης στα μέσα ενημέρωση. Ένα παράδειγμα του τι γίνεται στη χώρα μου. Το κυβερνών κόμμα αρέσκεται να μιλά για διάλογο, για συμβιβασμό, για την ε, θέληση να επιτύχει αυτόν τον συμβιβασμό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ένα σωστό διάλογο, να φτάσεις σε ένα συμβασμό όταν μιλάς μόνος σου. Και αυτή τη στιγμή έτσι έχει η σύνθεση του Κοινοβουλίου της Πολωνίας. Ε, αν ε, δείτε τους ε, συμμετέχοντες από το Πολωνικό Κοινοβούλιο, είναι όλοι από το κυβερνόν κόμμα. Κανείς δεν είναι από την αντιπολίτευση. Και νομίζω πως αυτό αρκεί για να αποφασίσετε μόνοι σας και να κρίνετε το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε μια τέτοια κατάσταση όπου το κυβερνών κόμμα έχει καταλάβει δια της βίας, της ομής μάλιστα βίας, αυτό το βήμα διαλόγου. Και είναι ενδεικτικό το ότι απουσιάζει η πλήρη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεμπρετόν, Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα συντομία να πάρω το λόγο για να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο σήμερα και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους των εθνικών διαμεσολαβητών, των οποίων πραγματικά εκτίμησα τις παρεμβάσεις γιατί αναφέρθηκαν σε αυτά ζητήματα. Ποιος είναι ο απολογισμός. Δεν με εκπλήσουν τα όσα άκουσα. Οι διαμεσολαβητές έχουν περιορισμένα μέσα δράσης γιατί αφορούν, βασίζονται περισσότερο στην δύναμη της πυθούς και όχι στη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς δεν μπορούν να επιτύχουν το 100%. Ο ρόλος τους όμως είναι αρκετά αποτελεσματικός και για να εφαρμοστεί το εθνικό και το νοσιακό δίκαιο. Αυτό ισχύει στη Γαλλία για παράδειγμα ο είναι διαμεσολαβητής στη Γαλλία είναι αρκετά αποτελεσματικός. Διαπιστώνω επίσης ότι αυτό συμβαίνει και με τους ομιλητές που πήραν το λόγο. Κατάλαβα ότι οι διαμεσολαβητές στη ε, Σλοβακία, στη Φιλανδία και στην Πορτογαλία είναι αρκετά αποτελεσματικοί. Με δυσκολίες βέβαια. Παρ' όλα αυτά επιτυχάνουν ορισμένα αποτελέσματα. Συνεπώς οι παρεμβάσεις τους είναι ιδιαίτερα εξισορροπημένες. Αντίθετα, με εξέπληξε λιγάκι η παρέμβαση του εκπροσώπου από την Πολωνία που δυστυχώ αναχώρισε κανένα μία αναχώρησε. Έκανε μια παρέμβαση ιδιαίτερα ε, απεσιόδοξη κατά την άποψή μου. Έδωσε μια ε, μάλλον προκατηλημένη ε, αντίληψη. Το ένα παράδειγμα αφορά ένα ευαίσθητο θέμα που είναι η μετανάστευση θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι από την κάνει ένας διαμεσολαβητής να υποχρεώσει μια χώρα να σεβαστεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε θέματα ε, μετανάστευσης αν δεν θέλει να το κάνει. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα κυριαρχίας. Τι είναι η κυριαρχία? Θα ήθελα εν συντομία να δώσω έναν ορισμό. Δεν είναι μια σειρά από αρμοδιότητες που εδρεώνονται από από μία συνθήκη και μεταφέρονται σε ένα υπερεθνικό όργανο. Η κυριαρχία είναι αυτό που είχε ο Καρλ Σμιτ, ο Γερμανός φιλόσοφος. Η κυριαρχία έγκυται στο να μπορεί κανείς να αποφασίσει για την εξαίρεση. Είναι η, δυνατότητα να μπορεί να αρνηθεί κανείς να συμμορφωθεί με το δίκαιο γιατί έχουν, έχει σχέση με τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας του. Και ε, εδώ ε, είναι ένα θέμα μετεγκατάσταση ε, των μεταναστών. Και εκεί ακριβώς υπάρχει αυτή η αντίληψη κατασμήτε σε ό,τι αφορά την κυριαρχία. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η δική μου ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να κάνει κάποια παρατήρηση, κάποια ερώτηση. Αν όχι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ομιλητές. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το μήνυμα είναι ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μία πρόκληση και για τις εθνικές και για τις ενωσιακές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας.